Θα δώσω την κυρία Φόρτ σαν αρμόδια εισηγήτρια για μας. Να τη δώσω το λόγο να μας παρουσιάσει τις σκέψεις και μετά να συζητήσουμε παρακαλώ συνάδελφοι. Thank you very much, Chairman, and for your brief update on the situation. I have to admit my frustration. Για να σας ενημερώσω Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την απογοήτευσή μου. Δεν ήρθε σε επαφή ο εισηγητής νομίζω μόνο πολύ πρόσφατα, χτες το απόγευμα, οπότε δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο. Έχω την αίσθηση ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση Άλλε επιτροπέ είχαν ε, αποκλειστικέ αρμοδιότητε, ιδιαίτερα στον τομέα της ευθύνη και οι νομοθετικέ αυτέ ρυθμίσει πρέπει να επανεξεταστούν. γιατί η κάθε επιτροπή πρέπει να είναι υπεύθυνη για το νομοθετικό έργο το οποίο η ίδια παράγει εν πάση περιπτώσει. Προσεκλήθησαν όλοι στην ανεπίσημη ακρόαση την οποία οργανώσαμε την Τρίτη. Ευχαριστώ και τα μέλη συναδέλφους εδώ που ήταν παρόντες. Ένας από τους κοιόδης επίσης ήταν εκεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και να συμπεριλάβουμε όχι μόνο μέλη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά και όσο περισσότερα μέλη γίνεται από το Κοινοβούλιο γιατί το θέμα έχει τεράστια σημασία. Μιλάμε για την διασφάλιση προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αλλά αυτό που προκάλεσε, αν θέλετε, ε, την έκθεση αυτή ήταν το τρομερό ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού. Πραγματικά η διαδικασία που ακολούθησε ήταν μια διαδικασία που έβγαλε τη βιομηχανία από την κόλαση ουσιαστικά. Αυτό όμως δεν συγχωρεί κανέναν, δεν δίνει κανένα άλοθη για κανέναν. Υπήρξαν τρομερά προβλήματα στη βιομηχανική αυτή δραστηριότητα και σε επίπεδο προσωπικού και σε επίπεδο διαδικαστικό και σε επίπεδο ασφάλειας από πλευράς των επιχειρήσεων χρηστών και ε, της ρυθμιστικής αρχής όπως επίσης και ενός νομοθετικού σώματος που θα το χαρακτήριζα οκνηρό. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα και για την βιομηχανία και για τις ρυθμιστικές αρχές και για τους νομοθέτες που και εμείς οι ίδιοι εδώ παίζουμε κάποιο ρόλο να επαναφέρουμε τα πράγματα σε καλύτερο επίπεδο. Άκουσα το καθεστώς το οποίο ισχύει στα δικά μας ύδατα, στα πιο όρημα σε επίπεδο βιομηχανικής δραστηριότητας όπως η Βόρεια Θάλασσα αν είχαν χρησιμοποιηθεί τα συστήματα αυτά στην, στην περίπτωση του κόλπου του Μεξικού, η τραγωδία δεν θα είχε ίσως συμβεί καν. Αν πάρουμε κανείς λοιπόν το ρυθμιστικό καθεστώς, το νομοθετικό καθεστώς και το προσαρτήσουμε αν θέλετε σε, έναν, σε μια ρυθμιστική αρχή η οποία να είναι πραγματικά ισχυρή και εν γνώση του θέματος τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους αυτής της δραστηριότητα και ε, να αποκλείσουμε ουσιαστικά τέτοιου είδους πιθανότητες για τα ευρωπαϊκά ύδατα. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι οι ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνονται από τρίτους ελεγκτές, δηλαδή ανεξάρτητους ελεγκτές, ελεγκτικές αρχές αυτό ισχύει για, σε κάποιες χώρες, όχι όμως σε άλλες, οπότε σε αυτή την περίπτωση τίθεται το θέμα της χρήσης της βέλτιστης πρακτικής. Την Τρίτη ζητήσαμε επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συναντηθεί με τις λεγόμενες αρχές του Φόρουμ της Βόρειας Θάλασσας. Αυτό το Φόρουμ της Βόρειας Θάλασσας περιλαμβάνει χώρες επίσης και από την Μεσόγειο, ας πούμε, Ιταλία από τη Μάλτα, Γάλλη και αυτό το οποίο συστήσαμε εμείς στα πλαίσια της πρότασης είναι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση και να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και κάτι τέτοιο θα πρέπει να ισχύσει και στη Μεσόγειο και όχι μόνο στη Βόρεια Θάλασσα και πρέπει να σας ενημερώσω ότι είναι σε φάση δημιουργίας τώρα ε, μια αρχή ε, για την ε, offshore άντληση πετρελαίου στη Μεσόγειο θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα βήμα προόδου. Η βασική προτεραιότητα βέβαια είναι να προλάβουμε μια τέτοια καταστροφή. Υπάρχουν ε, στην επιστολή η οποία έχει δοθεί στην διάσκεψη των Προέδρων, από την ε, διάσκεψη ε, των Προέδρων, υπάρχουν δύο λέξεις οι οποίες μου δημιουργούν ένα πρόβλημα. Αφορά την πολιτική προστασία, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Λέγεται εδώ ότι η, η διάρθρωση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί στα πλαίσια γενικότερα της ενίσχυσης της δυνατότητας αντίδρασης και ανταπόκρισης σε φυσικές καταστροφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη σε σχέση με τα πολιτικά μέσα, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για την πρόληψη των καταστροφών είτε φυσικών είτε όχι. Και αν με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ε, ρίχνουμε το βάρος της πρόληψης σε μια κοινοτική αρχή η οποία θα προλαμβάνει φυσικές καταστροφές ή καταστροφές του ΚΟΥΡ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα πρέπει να, να μην απεκδηθούμε των ευθυνών μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς σαν νομοθέτες διρίχνουμε τις ευθύνε στην πολιτική προστασία η οποία αν κάνει ό,τι μπορεί να κάνει δεν θα υπάρξουν καταστροφές. Πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές και πιο υπεύθυνοι. Πέραν αυτού πάντως υπάρχει ένα αφέστατος ρόλος σχετικά με την πολιτική προστασία. Υπάρχει επίσης ένα θέμα και σε σχέση με την πρόληψη. Στην περίπτωση του κόλπου του Μεξικού η αντίδραση από πλευρά των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση. Ελπίζω τέτοιες καταστάσεις να μην ε, ζήσουμε στη Βόρεια Θάλασσα Ελπίζω επίσης τα βήματα προόδου τα οποία έχουν επιτελεστεί στη Βόρεια Θάλασσα να περάσουν και στη Μεσόγειο. Υπάρχει λοιπόν κάποιος ρόλος και για την ΕΜΣΑ την Ένωση της Θάλασσας, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας της Θάλασσα. Νομίζω και εδώ υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στον τομέα της, ε, του καθαρισμού κυλίδων πετρελαίου στη θάλασσα. Ακούγοντάς τους για το αν τα τελευταία χρόνια τα πράγματα ήταν ικανοποιητικά ή αν απαιτούνται περισσότερες κτηριακές εγκαταστάσεις ή εν πάση περιπτώσει κάποιες ρυθμίσεις σε επίπεδο επιμελητιακό αυτό όμως είναι δευτερεύον. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, αν είχε υπάρ... ότι πρέπει να υπάρξει μια πιο συντονισμένη απόκριση στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοια προβλήματα. Αυτό που ακούσαμε επίσης την Τρίτη είναι ότι στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει μια κοιλίδα σε μια κλειστή θάλασσα όπως η Μεσόγειος, τότε οι περιβαλλοντικές συνέπειες θα είναι υψηλότατες. Οπότε η δυνατότητα άμεσης απόκρισης είναι κρίσιμη ιδιαίτερα αν <clears throat> δει κανεί και την απώλεια των δραστηριοτήτων οι οποίες θα επέλθουν σαν συνέπεια ιδιαίτερα σε κλειστά ύδατα. Ξέρουμε τι προβλήματα θα υπάρξουν στην ακτή της Βορείου Αφρικής σαν παράδειγμα. Γιατί αν μπορούμε να καλύψουμε και τα εδάφια αυτά, ακόμα και αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι προς όφελος όλων. Υπάρχει λοιπόν μια συνένεση και στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό το οποίο λέγω στην έκθεσή μου είναι ότι το θέμα της ασφάλειας δεν είναι θέμα ιδιοκτησίας, δεν είναι θέμα αποκλειστικό. Πρέπει να ρυθμίζονται τα θέματα της ανταλλαγής πληροφοριών όχι μόνο ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές. Υπάρχουν και μη επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες και υποχρεωτικές αναφορές και ανακοινώσει συμβάντων έτσι ώστε και οι υπόλοιπε χώρες να μπορέσουν να προετοιμαστούν για άμεση αντίδραση όταν υπάρχει ένα πρόβλημα ή όταν παραλίγο να υπάρξει ένα σοβαρό πρόβλημα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για την ελασχόληση στο παρελθόν και με την στρατηγική στη θάλασσα, την οδηγία πλαίσιο για τη στρατηγική στη θάλασσα. Αυτά είναι θέματα που συνδέονται με το συγκεκριμένο και θα πρέπει οι προτάσεις του στον τομέα αυτό να μην δημιουργούν κενά στην νομοθετική ρύθμιση την οποία συνολικά προτείνουμε. Εκεί τουλάχιστον που έχουμε και έχουν αυτοί οι αρμοδιότητες. Όπως είπα λοιπόν, πρώτον, θα πρέπει να έχουμε ένα καθεστώς ασφάλειας το οποίο να βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και το οποίο να βελτιούται συνεχώς. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή κατανομή και ανταλλαγή πληροφοριών, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές κάθε χώρα οι ρυθμιστικές αρχές. Τρίτον, θα πρέπει να έχουμε τα άμεστα καλύτερα τεχνικά μέσα για να προλαμβάνουμε την κλιμάκωση μιας καταστροφής να υπάρχει άμεσος καθαρισμός δηλαδή και τέλος πρέπει να υπάρχει άμεση αναφορά και ενημέρωση βασική προτεραιότητα κατ' εμές στον τομέα αυτό. <clears throat> Ξέρω ότι θα προσθεθούν και άλλα θέματα μέσω των τροπολογιών και θα ήθελα να ευχαριστήσω προκαταρκτικά τους συναδέλφους για αυτές. Νομίζω ότι ο Σκίνερ βιάζεται, οπότε ίσως να μπορούσατε πρόεδρε να του ζητήσετε το λόγο πρώτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας. Συνήθως Κίνερ έχει το λόγο, σε συζήτησε και πρώτος το λόγο, οπότε είναι εντάξει τα πράγματα. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ τη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές για την καλή μας συνεργασία. Ήμουνα βέβαια και στην ακρόαση της πρόλες. Άκουσα εκεί την κυρία Φόρτ. Τέθηκαν θέματα ζωτική σημασία που δείχνουν ότι έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε, όχι μόνο από την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού, αλλά και για την συμπεριφορά της βιομηχανίας σε αυτό το τομέα. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Όντως έχουν ε, ανέβει προδιαγραφές, παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια. Υπάρχουν ευθύνε από τις πρακτικές. Οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες είναι διατεθειμένες να κλείσουν την στρόφιγγα όταν διαπιστώνουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν εκατομμύρια, το ίδιο πρέπει να κάνουν όταν κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές ή το περιβάλλον. Το θέμα αυτό του πώς συμπεριφέρονται οι βιομηχανίες κάθε φορά είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε στο, περισσότερο στο βάθος. Το ότι βρίσκονται στα ανοιχτά οι εξέδρες εξόριξης έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε εύκολα να δράσουμε από τις ακτές. Εξαρτάται από τις καιρικέ συνθήκες. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι το πιο ανησυχητικό είναι η Μεσόγειος, η Βόρεια Θάλασσα και ίσως πρέπει να δούμε πάλι από την αρχή το θέμα της συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα. Γιατί βγήκε αυτό από την ακρόαση, όπως βγήκε επίσης και το ότι υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι με τον οποίο εφαρμόζονται οι πολιτικές. Ένα άλλο θέμα το οποίο κοιτάζουμε εδώ πολύ είναι η αντιμετώπιση, όχι μόνο η πρόληψη δηλαδή, αλλά όταν διαπιστώσουμε ότι η πρόληψη δεν έχει λειτουργήσει, όπως έγινε στον κόλπο του Μεξικού, πώς θα χτιστεί το κατάλληλο κέλυφος, τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τις συνέπειες. Πήρε δύο μήνες αυτό για να γίνει στον κόλπο του Μεξικού, ενώ δύο μέρες θα φτάνανε. Λόγω της γραφειοκρατίας, λόγω άλλων ε, πρακτικών δυσκολιών, χρειάστηκε πολύ περισσότερος χρόνος. Με την έκθεση αυτή πρέπει να πιέσουμε ώστε να μην ξαναπεράσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα δεν υπάρχει μία λύση που να κολλάει παντού όχι, υπάρχει ένα συγκεκριμένος τύπος που έχει φτιαχτεί και που ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό και πρέπει να πούμε ότι η βιομηχανία πρέπει να είναι έτοιμη εφόσον πρέπει να κλείσει η στρόφιγα, να βρουν έναν τρόπο να σταματάνε το πετρέλαιο και να είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να το κάνουν αυτό. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο η βιομηχανία, αλλά και ερευνητέ και επιστήμονες. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις που να επικαλύπτονται. Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές ρυθμίσεις που να είναι και αντιφατικές μεταξύ τους. Και μετά να καταλήξουμε σε μια λύση που να βασίζεται στον κατώτερο κοινό παρονομαστή. Αντίθετα, πρέπει να ενθαρρύνουμε την ιδέα για στενή συνεργασία. Να μην υπάρχουν διαφορές οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους αυτοί που πρέπει. Πρέπει να δούμε βέβαια και το, τις δαπάνες των χωρών. Αν χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκές, ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ε, δεν συμμετέχουν οι χώρες. Εγώ νομίζω ότι ξέροντας πώς κυκλοφοράει η μόλυνση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να δούμε πόσο πολύ μπορούμε να πιέσουμε, όχι μόνο εκεί που υπάρχει στενή συνεργασία ήδη. Η συνεργασία μέχρι τώρα πήγε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Καβάλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστώ τη Βίκη Φόρ για την πολύ καλή έκθεση και τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο εργάστηκε και να ευχαριστώ και τους κοιόδους συζητητές. Έχω τέσσερα σχόλια για την έκθεση αυτή. Σημεία που έχω ήδη συζητήσει με την εισηγήτρια και τους της Καταρχήν, η έκθεση αφορά κυρίως τον εξόριξη του πετρελαίου και θα πρέπει να είναι το κεντρικό θέμα και θα πρέπει να αναφέρουμε όμως και το αέριο, όπως και ο τίτλος αναφέρει το αέριο. Θα πρέπει να έχουμε και εμείς στο κείμενο την αναφορά στο φυσικό αέριο. Δεύτερο σημείο. Η έκθεση επικεντρώνεται στο ρόλο των κρατών μελών. Λείπει το ευρωπαϊκό επίπεδο Και βλέπουμε δυστυχώς όταν υπάρχουν μεγάλα δυστυχήματα ότι δεν υπάρχουν σύνορα και όρια και πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι' αυτό. Υπάρχει σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Κομισιόν, για την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Χρειαζόμαστε την εφαρμογή των βελτίστων πρακτικών. Χρειαζόμαστε επίσης διαφάνεια και ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να κοιτάξουμε παραδείγματο χάρη τι γίνεται στον τομέα των αερομεταφορών. Θα μπορούσε να είναι αυτό ένα καλό παράδειγμα συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν κάποιες ε, ομοιότητες και οι αεροπορικές μεταφορές εργάζονται πάρα πολύ καλά όσον αφορά αυτόν τον συντονισμό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Τρίτο σχόλιο. Τονίζει η έκθεση τον ρόλο της βιομηχανίας. Ναι, συνήθω βέβαια υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση, αλλά όσον αφορά του κανόνε, τον ορισμό των προτύπων, τον συντονισμό, όλα αυτά θα πρέπει να είναι θέματα για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ ότι αυτός ο βιομηχανικός κλάδος θα πρέπει να έχει την κύρια ευθύνη όσον αφορά την υπευθυνότητα και, τη και την χρηματοδότηση. Αλλά ε, η νομοθεσία και οι δαπάνες στον τομέα των... του συντονισμού θα πρέπει να είναι στα χέρια του δημοσίου τομέα. Υπάρχει λοιπόν ένας ρόλος για τον ιδιωτικό και ένας ρόλος για τον δημόσιο τομέα. Επίσης, η έκθεση επικεντρώνεται στην περιοχή της Βορειού Θάλασσας. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί, γιατί οι περισσότερες δραστηριότητες γίνονται εκεί. Υπάρχει ήδη αρκετή εμπειρία του North Sea Authority ε, Forum και αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι αυτές οι εμπειρίες, οι βέλτικες Βέλτισε πρακτικές και καλή νομοθεσία θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλου τομείς όπως στην Μεσόγειο, στην Μαύρη Θάλασσα και στην Βαλτική. Και δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε ευρωπαϊκές περιοχές, αλλά να δούμε και τι γίνεται στις γειτονικέ περιοχές. Παραδείγματο χάρη να γίνει κάτι στην ε, νότια όχθη της Μεσογείου θα έχει επιπτώσεις σε κράτη-μέλη. Θα ήθελα να πιστώ σε προσοχή σας στο σημείο 31 επίσης, όπου λέγεται ότι οι εταιρείε που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται να έχουν το ίδια πρότυπα όταν εργαστούν εκτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank Um, I too would like to thank Vicky Ford very much um, for the work that she's done on this and also. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Δίκη ε, και για την ακρόαση. Όσοι παρευρεθήκαμε σε αυτήν, ε, βρήκαμε ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσο ακούσαμε. Συμφωνώ πολύ με την θεμελιώδη προσέγγιση της κυρίας Φόρτ όσον αφορά την ασφάλεια. Είναι όντως πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, στέρες ε, βάσεις και ρήτρε για την ε, ασφάλεια. Πάνω σε αυτό μπορούμε να χτίσουμε παραπάνω και να το επεκτείνουμε κάπως. Πάντως υπάρχουν τρία σημεία στα οποία θα ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται πραγματικά με τις υψηλές προδιαγραφές και τις βέλτιστες πρακτικές. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κενό. Είναι πολύ καλή έκθεση εκεί που επιμένει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δουν ποιε είναι οι βέλτιστες πρακτικές, αλλά εκεί σταματάει. Και δεν λέει ότι πρέπει να επιμείνουμε, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει μία χώρα ή μία επιχείρηση η οποία παρά τις πληροφορίες που θα έχει, που θα κυκλοφορούν λοιπά, για κάποιο λόγο δεν θα τηρεί και θα σέβεται αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Και αυτό με ενοχλεί. Γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά όλα αυτά που λέει η Βίκη και οι ανησυχίες που εκφράζει όσον αφορά τον έλεγχο των ελεκτών και τα λοιπά, ότι μπορεί αυτό να μην βοηθάει αλλά θα ήθελα να ακούσω και κάτι για τον όφηση τσοροφόρουμ. Θέλω να μάθω περισσότερα για το μήπως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλες γεωγραφικές περιοχές, η Μεσόγειος για παράδειγμα. Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίσουμε την εφαρμογή υψηλών επιπέδων ασφάλειας και εφαρμογή βέλτιστων ε, πρακτικών εφόσον οι ελεγκτές ε, μαζί δρούν. Επειδή υπάρχει και προηγούμενο. Η κυρία Πιλέρτε Καστίγιο το βάζει και στην οδηγία για το Telecoms όταν αποφασίζουμε για ένα σώμα ρυθμιστών αντί για έναν οργανισμό της Επιτροπής με ενδιαφέρει πολύ μια τέτοια δυνατότητα. Ίσως ναι, γιατί έτσι ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ασφάλεια. Στην ε, ακρόαση διαπίστωσα ότι υπήρχε κάποια έλλειψη ενθουσιασμού. Εγώ νομίζω ότι γίνεται όμως και πρέπει να φροντίσουμε να γίνει. Η λύση ίσως είναι να ενισχύσουμε τον ρόλο των ίδιων των ρυθμιστών. Αυτό θα βοηθήσει και στην ανταλλαγή πληροφοριών, που γίνεται καλά σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν γίνεται καλά ε, μεταξύ ρυθμιστών από διαφορετικές χώρες, όπως εντοπίζει και η Βίκη. Αυτή είναι η δυναμία. Αυτό ήταν το ένα. Δεύτερον, για το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχουν κενά που έχουν να κάνουν με την ευθύνη η σχετική οδηγία για την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον δεν είναι αρκετά σαφής και το πεδίο εφαρμογή της θα έπρεπε να διευρυνθεί. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι υπεύθυνο για την άμεση, την έμεση ζημιά, για το ποιο πληρώνει. Και όπω είπε και η συγκήτρια, αν υπάρξει διαρροή πετρελαίου πιο κοντά στις ακτές θα έχουμε μεγαλύτερο ακόμα πρόβλημα από ό,τι είχαμε τώρα που έγινε στα νυχτά της θάλασσας. Και πώς θα ξέρουμε τώρα τι κάνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ύδατα πέρα από τα ευρωπαϊκά. Υπάρχει άποψη που λέει δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να το ψάξει, να δει τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως, αν βρισκόμαστε εκτός ευρωπαϊκών υδάτων, να μην πρέπει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να τηρούν ακριβώς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά καλό θα ήταν, γιατί εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε όπου και αν βρουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, λίγο πολύ να τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που ισχύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Φόρτ, κυρίως για το ανοιχτό πνεύμα που επέδειξε και που δέχτηκε κοινέ τροπολογίε. Έχω τέσσερα σημεία. Πρόληψη, αμοιβαιότητα, συνεργασία, έλεγχος και ευθύνη. Αναφέρθηκαν σε αυτά λίγο πολύ και οι προλαλήσαντες. Για το πρώτο, το ατύχημα της Φουκοσίμα και το ατύχημα στο Μεξικό, στον κόλπο του Μεξικού. Εδώ υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ των δύο αυτών ατυχημάτων. Δηλαδή, εφαρμόζουμε μια ιδιαίτερα περίπλοκη τεχνολογία και διαπιστώνουμε στον κόλπο του Μεξικού ότι δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε μια εξόριξη που δεν πάει καλά και στη Βουκουσίμα όταν και εκεί υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα ψήξης δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, ακόμα δεν ξέρουμε. Άρα πρέπει να επιμείνουμε πολύ στο θέμα της πρόληψης και της αξιολόγησης του κινδύνου. Αυτό που μας εκπλήσει είναι ότι έγιναν πολλές εξορίξεις, έγιναν πολλά τέτοια ατυχήματα και τι κάναμε. Δεν κάνουμε τα πάντα για να μπορούμε να προλάβουμε τα ατυχήματα. Δεν κάνουμε τα πάντα από πλευρά τεχνολογία. Ε, λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όλε οι επιχειρήσει πρέπει να επενδύσουν, να δώσουν χρήματα δηλαδή, ώστε να υπάρχει λύση σε περίπτωση ατυχήματο. Στην περίπτωση του κόλφου του Μεξικού εννοείται, αλλά βέβαια και για τα πυρηνικά. Για την αμοιβαιότητα και τη συνεργασία τώρα. Μίλησαν γι' αυτό κάποιοι σκιώδεις. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε εμπειρίες η κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της εμπειρίες. Δεν υπάρχει όμως κάποια δομή για να συγκεντρώνονται όλες αυτές οι εμπειρίες και να τις ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Έρχομαι τώρα στον έλεγχο. Για μένα η ΕΜΣΑ ευχαρίστως να έχει παραπάνω προνόμια, αλλά αυτά που λέει η κυρία Όλ δεν μου αφήνουν αδιάφοροι ότι ίσως πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας των ελεγκτών για να τηρούνται κάποιες στάνταρ ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για τελειώς τι νόημα έχει. Και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Όταν ο κύριος Σότιγκερ ζήτησε να γίνουν ε, δοκιμές αντοχής stress test και να πάει ένα σώμα ειδικών να ελέγξει όλα τα πυρηνικά εργοστάσια, ε, οι ευρωπαϊκές χώρες τι είπαν, είπαν όχι. Μεταξύ άλλων και η Γαλλία και η Αγγλία. Αν όμως γίνει ένα τύχημα, ένα ραδιανεργό σύννεφο δεν ε, έχει σύνορα, ούτε η μόλυνση της θάλασσας. Γι' αυτό και εγώ θέλω να υπάρχει σώμα ελεκτών που να πηγαίνει και να ελέγχει πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις, αν ανταποκρίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που θα έχουμε, γιατί οι κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλοι σε περίπτωση ατυχήματο. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος για την ευθύνη. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Όταν ε, κάνει σε μια επιχείρηση, και σε μεσαίο βάθος, γιατί και εκεί γίνονται ατυχήματα, να υπάρχει μια ευθύνη για το περιβάλλον. Και όσον αφορά τις αποζημιώσεις, να λαμβάνετε υπόψη ότι αποζημιώνουν και κάθε ζημιά στο περιβάλλον, σε περίπτωση κοιλίδας, πετρολοκυλίδας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συναδελφοί, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και το ρολόι, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στι μερικέ διάταξει. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το λόγο αυτή των τη συζήτηση μέχρι τώρα. Μπορούσα να μακρηγορήσουν κάπω περισσότερο. Τώρα θα έλεγα δύο λεπτά ο καθένα. Παύλο υπήρχε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε τον ε, επικεφαλή τη Αμερικανική Υπηρεσία, ε, τον κύριο Πεσό και ε, τον κύριο Βέζαντ και μας παρουσίασαν δυστυχήματα σε πλατφόρμες εξόρυξης ε, θα ήθελα αυτή η έκθεση να ενσωματωθεί στη δική μας έκθεση γιατί καταδεικνύει ποια είναι η δυνατή ανάλυση των στραλμάτων προηγουμένω, πριν γίνει δηλαδή αυτό το στοίχημα. Και δεν είναι το μόνο το πρόβλημα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και πυρηνικά ε, δυστυχήματα μας απειλούν και γι' αυτό θα πρέπει και εκεί να έχουμε έγκαιρα συστήματα ασφαλείας. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρος. Ο κύριος Γκίρεκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω με τις αρμοδιότητες. Θα πρέπει νομίζω να εξεταστεί αυτό το θέμα. Γιατί ξέρουμε πού μας οδηγούν όλα αυτά έχοντας υπόψη μας τι έγινε στην Καραϊβική. Θα πρέπει να έχουμε νέα τεχνικά πρότυπα λοιπόν. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν κάθε εξόριξη να προστατεύεται. Και να υπάρχουν επίσης και οι δυνατότητα ε, έτοιμα, θα έλεγα, τα καπάκια, αν μπορούμε να το ονομάσουμε, έτσι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση δυστυχήματο. Να μην τα ψάχνουμε εκείνη την ώρα δηλαδή. Τώρα βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρά πρότυπα όχι μόνο στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε στη Βαλτική, στην Βόρειο Θάλασσα. Μην ξεχνάμε και την Κασπία όμως, όπου γίνονται εξορίξεις και αναζήτηση πετρελαίου. Τα πρότυπα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προσποιηθούν και σε αυτές τις περιοχές. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να δίνουμε άδειε εξόριξη σε εταιρείε που δεν ακολουθούν τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, δεν συμφωνώ. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει τόσα πράγματα η ΕΠΟΠΗ που μπορεί να μιλήσει για την παστερίωση των τυριών, που μπορεί να συζητήσει για την ποιότητα των εξατμίσεων των αυτοκινήτων, που συζητάει για την σήμανση των ε, προϊόντων ε, των ηλεκτρικών στα ψυγεία, δεν μπορεί να επιβάλλει προδιαγραφές που να προστατεύουν τους πολίτες της σε κάθε περίπτωση. Μα τι πράγματα είναι αυτά. κάτι που θα κραγεί στη θάλασσα. Τι νομίζουμε, ότι μόλις γύρω από την πλατφόρμα θα μολύνει τη θάλασσα. Αν όμω γινόταν κάτι τέτοιο σε μια βρετανική επιχείρηση σε άλλες χώρες, τι θα γίνει. Τι θα απαντήσει στους πολίτες. Δίνουμε άδειε κλπ. κλπ. Λέει εδώ και ότι αυτό εξαρτάται μόνο από τα κράτη-μέλη. Ή διαβάζω αλλού για τους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ένα ελεκτικό σώμα δεν προσφέρει πρόσθετη αξία. Ή λέμε εδώ ότι η βιομηχανία έχει τον πρώτο ρόλο. Μα πρόεδρε, από πού και ως πού. Η οδηγία σε Βέζο 2. Για θυμηθείτε την, την παρακάμπτουμε. Γιατί για να μην ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα, τι κάναμε. Μειώσαμε το μέγεθος και τις ποσότητες αλλά κυρίες και κύριοι μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά κυκλοφορούν επικίνδυνα προϊόντα στις γειτονιές σας το βράδυ. Θέλω λοιπόν να είναι καλά ενημερωμένοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θέλω να, υπάρχει, να υπάρχουν υψηλά, υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και η βιομηχανία και η παραγωγή να υποχρεώνονται να τηρούν τα πρότυπα ασφάλειας. Και αυτό είναι υπέρ όλων και των μισθωτών και όλων των πολιτών δεν πρέπει η ελευθερία των μεν να πλήττει την ελευθερία των άλλων. Και αυτό γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα σύντομα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Πάνεκ ή κάποιον άλλον τέλο πάντων. Κανένα δεν είναι παρόν από την Κομισιόν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πρόεδρε και καλημέρα σας. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση που παρουσίασε και για τη συμμετοχή της σε διάφορες αψεκδηλώσεις που οργανώσαμε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτού του είδους την συζήτηση στο κοινοβούλιο είτε αυτό καταλήξει τώρα σε μια έκθεση ή σε κάποια άλλου τύπου έγγραφο δεν είναι δικό, δικό μας θέμα αλλά μας άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση και ότι υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ των μελών της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου φαντάζομαι για τα διάφορα αυτά θέματα. Αυτό για μας είναι πολύ ενθαρρυντικό. Βλέπουμε τώρα τους ε, κυρίους και κυρίες βουλευτές να αντιμετωπίζουν ακριβώς τα θέματα που είχαμε εμείς ορίσει στην έκθεσή μας τον Οκτώβριο. Υπάρχει λοιπόν φαίνεται σημαντική σύγκληση μεταξύ αυτών που θεωρεί η Κομισιόν και αυτών που θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να γίνουν. <clears throat> Θα μπορούσα να συμφωνήσω το κείμενο ως προτείνεται ε, ότι κάνει μια αναλυτική περιγραφή τη ε, της κατάστασης και κατάδειξη των προβλημάτων και δεν παρουσιάζει λύσεις, αλλά αυτό για μας δεν είναι πρόβλημα. Εμείς ήδη προτείναμε κάποιες λύσεις για τα προβλήματα που τα βλέπουμε και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί σας για το κατά πόσο οι λύσεις αυτές είναι οι κατάλληλες. Επίσης υπάρχει μεγάλος αριθμός αν έχει πλειοψηφία μελών που ζητούν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση στην λύση που θα εξευρεθεί. Αυτό το υποστηρίζουμε. Ταυτόχρονα βέβαια Θέλουμε ε, να μην ξεχνάμε τα θέματα της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παρέμβει μόνο εκεί που μπορεί να προσθέσει σε αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη ή οι διάφορες περιφέρειες. Μέχρι στιγμής ήταν φιλόδοξη τα θέματα, πολύ επίκαιρα. Υπάρχουν διάφορα τομείς όπου μπορούν να αλλάξει η αντιμετώπιση αλλά αυτό που μας παρουσίασε η βιομηχανία και σας είπα ότι δεν ήθελαν οι βιομηχανικοί κλάδοι να μας ε, ε, παρουσιάσουν ξεκάθαρα τις ε, προτάσεις τους και τα συμπεράσματά τους. Αυτά τα συμπεράσματα καταδεικνύουν και τα όρια μέχρι τα οποία μπορούν να συμβάλλει ο κλάδος. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες, αλλά μας είπε ότι ε, υπάρχει ένα περιορισμό όσον αφορά την ευθύνη. Εδώ πραγματικά πρέπει να δράσουν οι δημόσιες αρχές και είναι μεμονωμένα μεμενες για την αριστεία αλλά δεν μπορεί να είναι να πάρουν μια εγγύηση ότι οποιαδήποτε μονάδα, οποιαδήποτε επιχείρηση με την οποία έχει σε επαφή κανένας μπορεί πραγματικά να υποσχεθεί πλήρη ε, ε, πλήρη σύγκληση προς τα πρότυπα αυτά και ο κλάδος, ο κλάδος, το συνολικό όργανο δεν μπορεί βέβαια να αναλάβει ευθύνη για όλους. Οι θέσιμες τεχνολογίες και οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει όμως να είναι το πρότυπο όχι μόνο για, τους καλύτερους, ε, για τις καλύτερες επιχειρήσεις αλλά θα πρέπει να είναι το πρότυπο για όλο τον κλάδο. Κατά πόσο θα υπάρχει μια επιτροπή ε, ελεγκτών ή αν θα περάσει από την νομοθεσία ως έχει, δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το δούμε. και ελπίζουμε ότι θα αναπτύξουμε από κοινού μέχρι το καλοκαίρι τις πρώτες απαντήσεις, τις πρώτες λύσεις για να σας υποβάλουμε τις σχετικές προτάσεις. Ξέρω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο, Πρόεδρε, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά είναι σαφές ότι δεν θα μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα κατά πόσο θα παρέμβαση ή πρόληψη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και τα δύο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ισχυροί όσον αφορά την πρόληψη, να Ελεγχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα βιομηχανικό τομέα και η βιομηχανία παντού είναι ένα τομέα στον οποίο υπάρχει κίνδυνο. Πρέπει να ελεγχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο αυτό, αλλά υπάρχει ο κίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε από τον υστέρων ε, μηχανισμού παρέμβαση ότι εάν συμβεί κάτι να ελεγχιστοποιήσουμε τι ε, αρνητικέ επιπτώσει. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ υποκοδηματική τώρα, πολύ θετική και θα αποκομίσουμε διδάγματα από τη συζήτηση που θα συμπεριλάβουμε στη δική μας έκθεση. Θα σας ευχαριστώ. Η κυρία Φόρτ θέλει το λόγο ως συζήτητρια να το κληρώσει. Σας ευχαριστώ για όλα, για τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να σας καλύψω. Ας διευκρινίσουμε για το τι συζητάμε. δεν σημαίνει τεχνικά ότι όλη η, η άντληση από υψηλά βάθη γίνεται με υψηλή πίεση και η άντληση από χαμηλά βάθη, από ρηχά γίνεται με χαμηλή πίεση. Αυτό δεν, είναι, ε, ε, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Ας ε, υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αντληθεί το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, τα πράγματα από εκεί και πέρα σε επίπεδο τεχνικό και σε επίπεδο ασφάλειας διευκολύνονται. Για τα σχόλια του Σκίνερ θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να μην καταλήξουμε στο να μετριάσουμε τα επίπεδα ασφαλείας λόγω των επικαλύψεων στις ε, ρυθμίσεις θα πρέπει να αυξήσουμε την ποιότητα και όχι να υιοθετήσουμε τον χαμηλότερο κοινό παραδεσμα... παρανομαστή. Θα πρέπει να έχουμε τα τεχνικά μέσα που να διακόπτουν την άντληση το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχουν τέτοια συστήματα στην Ευρώπη σε λειτουργία και υπάρχει κι άλλο ένα σύστημα το οποίο σταματά την άντληση του πετρελαίου το οποίο έχει παραγγελθεί από την βιομηχανία και θα πρέπει τέτοιου είδους τεχνικοί εξοπλισμοί να υπάρχουν και στη Μεσόγειο και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο η ευθύνη αυτή για, την τοπική, για τον τοπικό περιορισμό ε, και για την τοπική διακοπή άντλησης ε, να μπορεί να γίνει με τα μέσα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτός είναι ο πιο σωστός δρόμος. Οι επιτόπου τεχνικοί υπεύθυνοι θα πρέπει να μπορούν να πάρουν την απόφαση αυτή, να κλείσουν δηλαδή ουσιαστικά το πηγάδι άντλησης ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι η βέλτιστη πρακτική και υπάρχει, είναι διαθέσιμη. Υπάρχουν διαφορές και μικρότερα προβλήματα ανάμεσα ε, στο φυσικό αέριο από ό,τι στο πετρέλαιο. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι το πετρέλαιο. Προφανώ και πρέπει να υπάρξει συντονισμό όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανάμεσα σε όλες τι εταιρείε που ε, επιχειρούν στο ίδιο πεδίο. Και εδώ η ΕΜΣΑ θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Συμφωνώ με τη Φιώνα σε σχέση με τον ρόλο τον οποίο μπορούν να παίξουν. Έχουν εκφράσει κάποιες διακδικήσεις πολύ συγκεκριμένες θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα πλωτά μέσα τα οποία χρησιμοποιούν είναι κατάλληλα επίσης και για την άντληση φυσικού αερίου και όχι μόνο για τις καταστροφές και τα ναυάγια των πλοίων, των πετρελαιοφόρων. Και εφόσον δεν υπάρχει επιτόπου ένα μηχάνημα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προβλέπεται η γρήγορη μετακίνησή του. Εφαρμόζεται η αρχή βέβαια του όποιο μολύνει πληρώνει, αλλά παρόλα αυτά η νομοθεσία δεν εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την αρχή. Αυτό το συγκεκριμένο θέμα λοιπόν πρέπει να επανεξεταστεί γιατί εντάσσεται στις αρμοδιότητες Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τα σχόλια της Φιώνα σχετικά με τις ανάγκες στο δημόσιο τομέα να ανταποκρίνεται σε κανόνες ασφαλείας. Τε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη ρύθμιση σε συνεργασία με τον νομοθέτη και αυτό το οποίο επίσης χρειάζεται είναι η ανεξάρτητη επίσης αρχή όταν υπάρχει δυνατότητα διασφάλισης της ελευθερίας του ελεγκτή έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όταν μια φυγατρική εταιρεία της συγκεκριμένη επιχείρησης αναλαμβάνει τον έλεγχο προφανώς δεν μιλάμε για αντικειμενική κρίση. Εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν τις διαδικασίες με τις κατάλληλες αποφάσεις. Υπάρχει ένα θέμα έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης ένα από τα μαθήματα που πήραμε από τι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν ότι είχαν ρυθμιστικέ αρχές αλλά δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένοι, δεν είχαν τη σωστή εμπειρία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχει σχημασία η σχέση ανάμεσα στην επιχείρηση και τη ρυθμιστική αρχή να βασίζεται στην αρχή του σεβασμού. Και αυτό απαιτεί ε, εμπειρία, απαιτεί εκπαίδευση και από πλευρά τη δημόσια ελεγκτική αρχή. Αυτό το διαπιστώσαμε και στα πλαίσια του φόρουμ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων στα ίδια επίπεδα ασφαλείας. Αυτό πράγματι θα θέλαμε σε παγκόσμιο επίπεδο να συμβαίνει. Όλες οι ε, αντλητικές δραστηριότητες να γίνονται με υψηλά επίπεδα ασφαλείας. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο αυτό βέβαια γιατί σε ορισμένες περιοχές ε, δεν υπάρχουν ισχυρά συστήματα ε, ανεξαρτήτου ελέγχου. Σαν παράδειγμα, στη βόρεια Αφρική, στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, η ρυθμιστική αρχή είναι οι εθνικές εταιρείες παραγωγής πετρελαίου. Οπότε εκεί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και δεν διακρίνονται οι εταιρείες αυτές από το πνεύμα ανεξαρτησίας τους, από την εξουσία. Προφανώ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την κοινοτική νομοθεσία σε όλου, αλλά πρέπει να υπάρξει βελτίωση και στι υπόλοιπε περιοχέ, Πράγματι για την ανταλλαγή πληροφοριών και το συνδυασμό των πληροφοριών και την καλύτερη χρήση του. υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν δομές συγκέντρωσης των πληροφοριών και της σωστής χρήσης τους, αλλά οι δομές αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, δεν είναι δεσμευτικές και δεν είναι τόσο λειτουργικές όσο θα θέλαμε να είναι σε σχέση με την χρηματοδότηση των μηχανισμών περιορισμού της μόλυνσης και περιορισμού και μετρίασης των συνεπειών της. Προφανώς υπάρχει εδώ ένα θέμα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες επενδύσεις σχετικά με τις πρακτικές περιορισμού της άντλησης ή μάλλον διακοπής της άντλησης μέσω χρήσης εκρηκτικών. Υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και σε αυτό το τομέα αλλά μένει ακόμα πολλά να γίνουν. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο τη ημερησίας διάταξης. Ε, θα πρέπει να αποφασιστεί το θέμα που σα είπα στη διάσταση προέδρων. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 έως 7, πολιτική για το ραδιοφάσμα. Ο Γκούνορ Χοϊπμαν έχει το λόγο και να προχωρήσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους κοιόδης για τις ε, διάφορες ε, τροπολογίες που είναι όλες επικοδημητικές και όλες τονίζουν την σημασία του θέματος. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μια σειρά συμβιβασμών που ασχολούνται με αυτές τις ανησυχίες χωρίς να εγκαταλείψουμε το βασικό μας στόχο. Θα ήθελα πριν περάσω στη συζήτηση των διαφόρων τροπολογιών να τονίσω, Πρόεδρε, τι αφορά το θέμα αυτό. Στη δεκαετία του 90 η Ευρώπη ήταν η επικεφαλής όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία. Χάσαμε μετά τον ηγετικό αυτό ρόλο. Και βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η εξέλιξη του διαδικτύου και του δικτύου ευρύου φάσματος όχι μόνο για τον ίδιο τον κλάδο αλλά με επιπτώσεις στην εξέλιξη της κοινωνίας της ίδιας από οικονομικής πλευράς, πολιτιστικής πλευράς και πολιτικής πλευράς. Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα στον στόχο μας να ε, καταστήσουμε την Ευρώπη μια ηγετική οικονομία παγκόσμια. Και είπα Λιστάκης, όταν συζητάγαμε την έκθεση αυτή στο παρελθόν, Πρόεδρε. Εάν θέλουμε να παίζουμε τον ηγετικό ρόλο, θα πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. αν θέλουμε να είμαστε η τρίτη και όχι οι πρώτη, να πάρουμε την απόφαση να είμαστε η τρίτη. Αλλά δεν είδα πολλούς να θέλουν να διαλέξουμε να είμαστε η τρίτη. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλες και όλες οι συζητήσεις που είχαμε συμβάλλουν στις προσπάθειες να αδράξουμε τις καλύτερες ε, δυνατότητες για να παίξουμε τον ηγετικό αυτό ρόλο. Σε στο μέσο έχουμε φορέ απόψει, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε τις αλλαγές. Δεν μπορούμε να βασιστούμε δηλαδή στο τι γινόταν στο παρελθόν αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές. Και μπορούμε με ε, να καλύψουμε όλες τις ενισχύσεις που έχουν εκφραστεί. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα θέματα που είναι ουσιαστικά στη συζήτηση. Το πρώτο είναι η λεγότερη σύγκρουση μεταξύ της τηλεόρασης και των νέων τεχνολογιών, των νέων υπηρεσιών. Συζήτηση μεταξύ των ε, σκιωδών καθίσαμε απόλυτα σαφές ότι αυτό δεν πρέπει να είναι μια σύγκρουση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες συντονισμού της τηλεόρασης ε, και των νέων υπηρεσιών. Μπορούμε να κρατήσουμε ε, την, ε, την τηλεόραση όσο έχει σήμερα. Ίσως χρειαστούμε κάποιες αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα θυσιάσουμε οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να είναι σαφές και θα εκφραστεί και στις διάφορες συμβαστικές τροπολογίες. Θα πρέπει να προσθέσουμε να καλύψουμε όλα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα εδώ και να είμαστε σοβαροί και να αντιμετωπίσουμε το θέμα με σεβασμό. Γιατί τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Χρειαζόμαστε και κοινέ λύσεις. Επιτρέψτε μου να περάσω στην κατάσταση της δεκαετίας του 90 όταν είχε την ηγεσία η Ευρώπη. Γιατί είχε συμβεί αυτό, για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί απελευθέρωσε τις αγορές τηλεπικοινωνιών. Και επίσης, γιατί είχαμε ένα κοινό πρότυπο DSN που έδωσε τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι αγωνιστική και στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Αυτό ήταν ουσιαστικό, στρατηγική σημασία. Και θα πρέπει νομίζω να σκεφτούμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να σεβαστούμε αυτό που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, ταυτόχρονα όμω να καταβάλουμε προσπάθειε, ούτω ώστε κάτω τη δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε εναρμόνιση και συντονισμό με στόχο να ανοίξουμε μια αγορά με πανευρωπαϊκές ευκαιρίες και υπηρεσίες πολλών ειδών. Εάν δεν θέλουμε να το κάνουμε, ας πάρουμε τη σχετική απόφαση. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένα θα θέλει να πάρει την απόφαση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε αυτά όλα να, να καθιστούν δυνατά. Μία σειρά τροπολογιών αναφέρονται στην ιδέα μιας νέας τεχνολογίας. Τις ε, χαιρετίζω και θα ενταχθούν στις διάφορες συμβαστικές λύσεις. Γιατί βέβαια χρειάζεται να ε, λάβουμε υπόψη μας την ε, εκμετάλλευση όλων των νέων δυνατοτήτων όλων των δυνατοτήτων και να είμαστε σίγουροι ότι μια τεχνολογία δεν παρεμβαίνει σε άλλες τεχνολογίες. Πολλά γίνονται στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να το τονίσουμε εμείς στην έκθεσή μας. Χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη και οι διακανονιστές να τα λάβουν αυτά υπόψη τους. Ένα άλλο θέμα είναι τι γίνεται όταν πρέπει κανένας να αναδιανύμει ή να μεταφέρει διάφορες υπηρεσίες μέσα στις πλαίσεις του φάσματος. Συμβαστικές λύσεις ε, προτείνουμε τη δυνατότητα ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν και μπορούν να φροντίσουν να είναι δυνατές αυτές οι μεταφορές χωρίς να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα για τις ισχυούσες υπηρεσίες. Εν ολίγης έχουμε κάπου 50 τροπολογίες κύριε Πρόεδρε. Εγώ ελπίζω να μπορέσω να τις καλύψω με τις 21 συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε σήμερα και θα σας ε, βοηθήσουμε έτσι για την ψηφοφορία, Πρόεδρε. Ταυτόχρονα όμως θα μας βοηθήσει εμάς όλους να διατηρήσουμε τον κοινό στόχο να έχουμε μια ισχυρή έκθεση και ισχυρή υποστήριξη της. Οι συζητήσεις μεταξύ των σχεδόν είναι πολλά υποσχόμενες μέχρι στιγμής. Να αναφερθώ λίγο στις λεπτομέρειες. Πολλοί από τους συναδέλφους ήθελαν να ε, συνδυάσουν τη συζήτηση για τους στόχους και για το έβρος ε, αυτό το χαιρετίζω και θα συμπεριληφθεί στις συμβαστικές τροπολογίες ε, υπαριθμών 1 και 2. Και εσείς μεταξύ άλλων πρόεδρε υποβάλλετε τη σχετική ε, πρόταση και χαίρομαι πάρα πολύ να μπορέσω να καλύψω τις προτάσεις σας. Όσον αφορά τις διακονιστικές αρχές και πώς θα εφαρμοστούν πώ θα εφαρμοστεί η διάκριση μεταξύ των διαφόρων τρόπων χρήση τη τεχνολογία. Είχαμε διάφορε τροπολογίε που προσπαθούν να παρουσιάσουν σύνδεση προ τη δέσμη τηλεπικοινωνιών. Και προσπαθούμε να βρούμε μια συμβαστική που θα είναι ικανοποιητική για όλου. Κατόπιν όσον αφορά τις, ε, ε, πολιτικές που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ε, λέμε για τον αριθμό των MHz που θα έχουμε μέχρι το 2015. Ορισμένοι τονίζουν τη σημασία και χαίρομαι ότι ορισμένοι συναδελφοί υποβάλλουν τροπολογίες που τονίζουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη στην Ευρώπη να έχουμε το μεγαλύτερο διαχείριτα, το μεγαλύτερο δυναμικό και θα το τονίσω ακόμα περισσότερο στη συμβαστική πρόταση. Επίσης όσον αφορά το άρθρο 3 αυτό που είναι σημαντικό είναι μια σειρά τροπολογιών από πολλές πολιτικές ομάδες που τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη διαφορετικές αρχές ε, της ε, ευρυζωνικής ε, προσφοράς στα διάφορα κράτη, στους διάφορους πολιτιστικές παραδόσεις. Να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι δεν ξεχνάμε αυτό που είναι σημαντικό σήμερα. Από την άλλη μεριά δεν εγκαταλείπουμε την ανάγκη μεταρρύθμισης για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για το μέλλον. Ανταγωνισμός. Ε, και εκεί έχουν υποβληθεί μια σειρά ε, τροπολογιών ισχυρότερε από αυτό που είχα προτείνει αρχικά και θα χαρώ πάρα πολύ να τι λάβω υπόψη μου γιατί αυτό είναι από τα κεντρικά θέματα. Δεν είναι στατικό το θέμα. Ο κλάδος αυτός εξελίσσεται και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι νέοι ε, ε, ε, επιχειρηματίες, νέοι λειτουργοί μπορούν να εισέλθουν στην αγορά αυτή και να παρουσιάσουν γλίγορες αλλαγές. Και αυτά βέβαια, Πρόεδρε, καταλήγουν σε αυτά που υπάρχουν στο άρθρο 6 όπου οι περισσότεροι συνάδελφοι υποστηρίζουν τον δικό μου στόχο να παραμείνουμε δηλαδή στην προθεσμία του 2013. Άλλοι προτείνουν κάτι το διαφορετικό, αλλά οι περισσότεροι από τους συναδέλφους εδώ είχαν τονίσει την ανάγκη να γίνει αυτό και ταυτόχρονα την ανάγκη να σεβαστούμε εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν ιστορικής μορφής ε, προβλήματα. Σοβιετική δηλαδή, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Λευκορωσία που μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα στη διαπραγμάτιση για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ε, ε α, αυτές τις συχνότητες. Προχωράμε λοιπόν συζήτηση μεταξύ των σκιωδών, ορίζοντας τους στόχους αλλά αναφερόμενοι και στους λόγους εξαίρεσης από τους στόχους αυτούς. Όσον αφορά άλλα τμήματα του φάσματος, υπήρχε μια ευρεία ε, συνένεση όσον αφορά την επιλευθέρωση του 2,3 και του 1,5 για να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή συνένεση. Και μετά έχουμε βέβαια το πολύ σημαντικό θέμα και ευαίσθητο θέμα των 700 του φάσματος των 700. Άλλοι δεν θέλουν να αναφέρεται, άλλοι θέλουν να αναφέρεται ακόμα περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Θα θυμόσαστε ότι εγώ στην έκθεσή μου προτείνω να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αναθεωρήσει και να προετοιμάσει τη σχετική συζήτηση. άκουσα διάφορες ομιλίες ε, πολιτικών ηγετών που λένε η αύριο αρχίζει σήμερα. Το έχουμε ακούσει όλοι νομίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ αληθές όταν αφορά τα φάσματα. Γιατί εάν το φάσμα των 700 πρόκειται να ανοίξει για τα κινητά, τα κινητές υπηρεσίες το 2016, όταν γίνει μια διεθνή τηλεδιάσκεψη, εμείς θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει το 2012 για την τελεδιάσκεψη αυτή για να μπορεί να τεθεί το θέμα στην ημερησία διάταξη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση τώρα ότι θα θέλουμε να φυγεί το θέμα. Και να πούμε ότι δεν συζητηθεί καθόλου αυτό το 2016 και θα να χάσουμε αυτή την ευκαιρία αυτό νομίζω ε, θα ήταν ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε καθόλου υπεύθυνοι. Αυτό που αναφέρεται σε ένα συμβιβασμό ε, που τυχαίνει ευρεία συνένεση νομίζω ότι θα αναθεωρήσουμε και θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να δράσει να θέσει το θέμα για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε δυνατότητα να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε λοιπόν μία απόφαση για τα 700, για το φάσμα των 700, αλλά θα πρέπει, δίνουμε στην, ε, στους εαυτούς μας τη δυνατότητα να δράσουμε στο μέλλον. Αυτός ο συμβασμός νομίζω θα τύχει ευρύτατης συνένεση. Σε γενικές γραμμές, Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα δουν ότι έχουν καλυφθεί οι ανησυχίες τους. Για τις παραδοσιακές υπηρεσίες και πώς θα αντισταθμιστούν. Ε, είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξιών από τη συνεργική πρόταση. Αυτό είναι πολύ καλό. Μέχρι τούτο, Πρόεδρε, έχουμε σαν στόχο να είμαστε οι πρώτοι. Ευχαριστώ. Jens Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Χακμά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χέπμαν για την πολύ πραγματιστική και ευέλικτη στάση που κράτησε στις διαπραγματεύσεις τους. Προσπαθήσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να λάβουμε υπόψη μας ε, τις πολλές τροπολογίες, ιδίως εκείνες που προέρχονται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, συγγνώμη, πολιτισμού. Είναι νομίζω σαφές ότι με την νομοθεσία αυτή για την πολιτική φάσματος έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Ε, μπορούμε να άρουμε πολλά εμπόδια αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε τολμηροί για να εξασφαλίσουμε έντονο λογιστό με πολλούς συμμετέχοντες. Πρέπει να φροντίσουμε οι καταναλωτές να έχουν τις καλύτερες δυνατές προσφορές, τις καλύτερες δυνατές τιμές, χωρίς να χρειαστεί να διακανονίσουμε τις τιμές αυτές. Θα πρέπει να δειχθούμε τολμηροί ούτως ώστε να πάρουμε τα σωστά και σημαντικά βήματα για το μέλλον. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα όμως ότι δισεκατομμύρια ευρώ διακυβεύονται με την νομοθεσία αυτή. Εάν δεν το ξέραμε στην αρχή της διαδικασίας, το ξέρουμε τώρα. Γιατί έχουμε συναντήσει όλοι πολλούς ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι μιλάω γερμανικά σήμερα έχει κάποιο λόγο. Ε, είδα έντονη δραστηριότητα γερμανικών λόμπι ε, και μου φαίνεται ότι εντάξει, μου αρέσει αυτό. Αλλά υπάρχει ένα τομέας στον οποίο ο κλάδος ε, ο πολιτιστικός στη Γερμανία σφάλει. Δηλαδή εκεί που δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του ανοίγματος νέας τεχνολογικής πλατφόρμας και την διατήρηση του περιεχομένου και του πολιτισμού. Λυπούμε. Δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να τεθεί αυτή η, η αντίφαση, γιατί ο πολιτισμός είναι ουδέτερος όσον αφορά την τεχνολογία. Μπαίνει από παντού. Και όσο πιο φτηνή είναι η δυνατότητα διάδοσης, τόσο πιο έντονη είναι η διάδοση του πολιτισμού αυτού. Εγώ θα πω στα μέλη της πολιτικής πολιτισμού ότι η πολιτιστική εξέλιξη δεν θα περιοριστεί με την νομοθεσία αυτή, αλλά θα ενδυναμωθεί. Όταν οι δημόσιες ε, εταιρείες ε, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης προσπαθούν να δώσουν την εντύπωση αυτή, διακυβεύεται κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχει η επιθυμία δια τήρησης του ρόλου θηρορού που παίζουν. Εγώ εδώ και 15 χρόνια ασχολούμαι έντονα με θέματα φάσματος. Ξέρω τι παιχνίδι παίζεται. Η επιθυμία να διατηρηθεί αυτός ο ρόλος θηρορού είναι κατανοητός. Νόμιμος θα έλεγα. Αλλά οι προϋποθέσεις είναι εσφαλμένες. Όταν βλέπουμε ότι στη μια ανθρωπολογία μετά την άλλη παρουσιάζεται μία αντίφαση μεταξύ της διατήρησης ε, του πολιτιστικού περιεχομένου και της προώθησης τεχνολογίας. Θα ήθελα να πω προς τον κύριο Χέκμαν σήμερα ότι εκτιμώ πάρα πολύ το ενδιαφέρον που δείχνει για το θέμα και την κατανόηση προς τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Βιομηχανίας, αλλά λυπούμε που ένα τόσο ραμπατικό έγγραφο βασίζεται σε εσφαλμένες προϋποθέσεις όσον αφορά αυτή την αντίφαση μεταξύ τεχνολογικής και πολιτιστικής εξέλιξης. Του αντίον. Η κατεύθυνση που ακολουθείτε ακόμα είναι σωστή. Σας παρακαλώ όμως να διατηρήσετε την κατεύθυνση αυτή. Χρειαζόμαστε ισχυρό ευρωπαϊκό ανταγωνισμό με τεχνολογική εξέλιξη, απελευθέρωση και κοινό ευρωπαϊκό πεδίο παιδείς. Αυτό θα το εκπληκτήσουν όλοι οι τελικοί χρήστες. Γιατί θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν σωστά για και από οικονομικούς, πολιτιστικούς και άλλους λόγους και ελπίζω να έχουμε τελικά ένα ισχυρό αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ρουμπίχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε νομίζω μια ιστορική ευκαιρία τώρα να περάσει ή να σκεφτούμε μάλλον πάνω στη μεταφορά αυτή προς τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ε, το ρόλο μας στο κοινοβούλιο, όπως και ε, μέχρι τώρα, είναι να δώσουμε μια εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα εθνικό θέμα, αλλά θα πρέπει να διακανονιστούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα υπερεθνικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2016 και ούτε να περιοριστούμε σε κάποια λίγα φάσματα. Άρα θα πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε αυτή την ευκαιρία ως Κοινοβούλιο. Και είναι σαφές ότι η εντολή αυτή ισχύει για τις εν λόγω προσφερόμενες ε, συχνότητες, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε ότι αν κάποιες συχνότητες δεν ε, χρησιμοποιούνται μπορούν να διατηθούν ας πούμε κάπου αλλού για την ε, τις υπηρεσίες ε, ε, σε περίπτωση καταστροφής ή άλλο που χρειάζονται μια δεύτερη συχνότητα και θα πρέπει σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα, σε ένα φάσμα συχνότητας να είναι δυνατή η ασφαλής επικοινωνία. Και όπως επιβεβαιώ αυτό θα μπορέσει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και θα πρέπει εδώ να κληθεί η Κομισιόν ξεκάθαρα να εξετάσει και αυτή την εντολή αυτή για να μπορέσουμε μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιών πρώτης ανάγκης και σε περίπτωση καταστροφής να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια στον κύριο Χόκμαρτ, τον συναδελφό μου, για την εκθεσή του και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να μας οδηγήσει στις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Το έκανα αυτό με πολύ ταλέντο. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τι περιλαμβάνεται τώρα και τι δεν περιλαμβάνεται σε αυτές. Πάντως, έχω να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις μετά από αυτά που τον άκουσα να λέει. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια τάση στους φορείς ε, κινητής ε, τηλεφωνίας για το φάσμα ορισμένοι και επικοινωνιών που ορισμένοι θέλουν να αποφύγουν το πολιτιστικό περιεχόμενο, άλλοι αντίθετα. Καταλαβαίνω την οπτική γωνία αυτών των δύο πλευρών, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να νιώθουν ότι απειλούνται όσοι πιέζονται από τα 700. Είπαμε ότι μπορούμε να το αλλάξουμε, να πετύχουμε ένα συμβιβασμό. Μην βιαζόμαστε πάντως να βγάλουμε τους φορείς από το φάσμα το οποίο χρησιμοποιούν τώρα. Μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος χρειάζεται περισσότερο φάσμα, θα το πάρει. Θεωρώ ότι παραβλέπουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσω της κοινοτομίας και της τεχνολογικής πρόοδου και ίσως να έχουμε ξεχάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Ίσως κάποιοι στις κινητές επικοινωνίες να μπορέσουν να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί και να μην χρειαστεί αυτό το εύρος. Υπάρχει και τηλεόραση και μην ξεχνάμε ότι παντού υπάρχει καινοτομία. Έχουμε παρακολουθήσει διάφορες παρουσιάσεις νέων τρόπων χρήσης της ευρυζωνικότητας και του περιεχομένου. Καταρχήν συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Ρούμπικ Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά κενά, λευκά ε, κενά στο, στην ευρυζωνικότητα που τα κρατάμε για διάφορες περιπτώσεις και για διάφορες αρχές. Πρέπει να δούμε λοιπόν με αυτές τις αρχές και με τα κράτη-μέλη ώστε να αιτιολογούν πώς χρησιμοποιούν την ε, ευρυζωνικότητα. Ποιοι θα πρέπει να κάνουν τον κόπο και να υποστούν τις αλλαγές. Γιατί να προστατεύουμε τον δημόσιο τομέα. Αν μη τι άλλο να τους ζητάμε να αιτιολογούν το πώς χρησιμοποιούν τις συχνότητες. Και το ξέρουν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μια τάση να ξέρουμε που πάντα χρήμα. Στη χώρα μου τουλάχιστον ισχύει αυτό όταν θέλουμε να κάνουμε περικοπές πρέπει να χρησιμοποιείτε τα χρήματα όσο γίνεται καλύτερα. Πολλοί μου γράφουν από την εκλογική μου περιφέρεια προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, κάτι τεχνικό, το οποίο δεν έχει λυθεί από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι οι παρεμβολές ανάμεσα στους φορείς του καλωδιακού και των κινητών ε, επικοινωνιών. Φαίνεται ότι υπάρχει παρεμβολή από τις κινητές επικοινωνίες. Δεν υπάρχει καμιά έτοιμη λύση. Χρειάζεται όμως συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και των ρυθμιστών για να λυθεί αυτό να βρεθεί κάποια λύση στην πράξη. Γιατί κανέναν δεν βοηθάει να υπάρχουν τέτοιες παρεμβολές στις συχνότητες τελικά ο καταναλωτής πλήττεται. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χόκμαρκ για την δουλειά που έχει κάνει και περιμένω και εγώ ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Λάμπερτς, ο κύριος... Λάμπερτς αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε Uh, like to... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κούναρ για την προσπάθεια που έκανε και για τις συμβιβαστικές τροπολογίες μια πολύ καλή δουλειά του και θα μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε αν όχι όλες τις περισσότερες. Να επαναλάβω αυτά που είπε ο για το ότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εκπομπές ε, ε, προτείνουν. Αυτοί που διαχειρίζονται την κινητή τηλεφωνία δεν είναι το α και το ω του μέλλοντος. Πολλοί πρέπει να διαχειριστούν τον χώρο αυτό του φάσματος. πρέπει να διασφαλίσουμε το δικαίωμα κάποιων επιχειρήσεων να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι ε, κοινή ιδιοκτησία, καθολικού τύπου ιδιοκτησία. Υπάρχουν ε, κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα και οι οποίες εκπέμπουν στο φάσμα συχνοτήτων και θα μπορούν να ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση με όλους τους άλλους. Δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο οι αρχές ή οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν σε ορισμένες επιχειρήσεις διαφορετική μεταχείριση από τις άλλες. Σχετικά τώρα με τις αποστολές κοινή ωφέλειας. Είναι προφανές ότι το σύνολο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό. Και εδώ ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες ειδικέ ρυθμίσεις για αυτό το τμήμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών, οι οποίες δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να την χάνουν κάποια επίπεδα προστασίας και ε, διασφαλισμένης πρόσβασης. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τα αναμειγνύουμε αυτά τα δύο. Δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την κοινή ωφέλεια η οποία είναι πολιτιστική μερικές φορές αλλά μερικές φορές είναι ε, απόλυτα εμπορική δραστηριότητα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ελεύθερη αγορά, υπάρχει ανταγωνισμός στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, έτσι λειτουργεί η αγορά. Και το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας. Εφόσον παρέχουν περιεχόμενο και εφόσον παρέχουν ενδιαφέροντα προϊόντα τα οποία πολλούνται τόσο το καλύτερο. Αν δεν το κάνουν αυτό θα αποτύχουν. <clears throat> Υπάρχει όμως ένα τμήμα του πολιτισμού το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι κοινή ωφέλεια, δεν είναι κάτι το οποίο θα ε, ε, προσφέρει κέρδη, χρήζει ενίσχυση και προστασία. Α κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα δύο. Αν τα αναμειγνύουμε αυτά τα δύο τότε φοβάμαι ότι θα έχουμε ανυπέρβλητα μπροστά μα προβλήματα. Σα ευχαριστώ. Εάν συμφωνείτε, έχοντα κατόπιν και το ρολόι και του νόμου που έχουν το επόμενο σημείο τη ερμηνεία διατάξη, θα ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτηση. Κανένα άλλο δεν έχει συζητήσει το λόγο ούτω ή άλλω. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τι 12 Απριλίου. Δεν υπάρχουν θέματα ανοιχτά ότι είναι ανοιχτό, θα το συμφωνήσουν οι συνάδελφοι μεταξύ τους επόμενες εβδομάδε. Ευχαριστώ αυτού που έχουν εργαστεί. Θα μου πρέπει να πάω στο επόμενο σημείο τώρα, στο θέμα τη καινοτομία. Και θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μέρκης. Σημείο 5. Thank you, Chairman. Um... Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει. 302. 8 γνωμοδοτήσεις επίσης από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα της καινοτομίας, της Ένωσης Καινοτομίας, μια που η καινοτομία είναι μια λέξη κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να να επιτευχθεί μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και να βγούμε από την ε, κρίση. Προσπαθώ να ετοιμάσω συμβαστικές τροπολογίες. Όσο επί το πλήστον νομίζω ότι συμφωνούμε για το πόσο μεγάλη σημασία έχει η καινοτομία και για το τι στοιχεία χρειαζόμαστε προκειμένου να την επιταχύνουμε και να την αντιναμώσουμε. Ε, Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα, πιστεύω ότι θα πετύχουμε συμφωνία. Κάποια σημεία όμως πρέπει να διευκρινιστούν παρετέρω. Πρέπει να βρούμε καλύτερη διατύπωση για αυτά ή έναν καλύτερο ορισμό ίσως του τι ακριβώ θέλουμε. Για παράδειγμα, υπάρχει το επιχειρίζεστε ε, σε αντιπαράθεση με τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Βλέπετε, σε αυτό το τρίγωνο ή το διαμάντι που το λέω εγώ, Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν στοιχεία κλειδί για την καινοτομία. Έτσι λοιπόν τα χρειαζόμαστε και τα μεν και τα δε. Εδώ δεν είναι σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε μια επιχειρηματική προσέγγιση. Χρειαζόμαστε τις επιχειρήσεις, αλλά χρειαζόμαστε και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε ο καθένας να έχει το δικό του ρόλο. Έπειτα υπάρχουν οι πολίτες από την μια μεριά και επιχειρήσεις από την άλλη. Και αυτό είναι ένα επίμαχο θέμα. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι έτσι. Δεν είναι σε αντιπαράθεση μεν με τους δε. Η επιχείρηση στο κάτω-κάτω τι είναι. Είναι ένας ε, ε, πολίτης ή μια ομάδα πολιτών οι οποίοι παράγουν κάτι. Ο πολίτης είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας και έχει πολλούς ρόλους, όπως ένας πολίτης σε μια δημοκρατία που έχει και υποχρεώσεις και καθήκοντα, αλλά μπορεί να είναι και υπάλληλο και επιχειρηματίας και ερευνητής ή πολιτικός. Συνεπώς, ένας πολίτης έχει ρόλο παντού, σε κάθε θέση. Η δημιουργικότητα λοιπόν, το επιχειρίζεστε, η περιέργεια που επιδεικνύει ο πολίτης είναι και το στοιχείο κλειδί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό πρέπει να δυναμώσουμε. Αυτό πρέπει να ενισχύσουμε. Αν έχουμε περιέργεια, αν έχουμε πολίτες που καινοτομούν, που κάνουν επιχειρήσεις, τότε θα πετύχουμε στην έρευνα, στο επιχειρίζεστε, στις κυβερνήσεις κτλ. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να βρω τη σωστή διατύπωση, την κατάλληλη διατύπωση για να το δείξω αυτό στην έκθεσή μου. Δεν πρόκειται για αντιπαράθεση των μεν με τους δε. Επίσης έχουμε την κοινωνική κοινοτομία και την οικονομική καινοτομία από την άλλη μεριά. Πρέπει να σα πω ότι πριν έρθω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα όλη μου τη ζωή, σε επιχειρήσει. Και ακόμα και αν είμαι στους σοσιαλιστές σήμερα, πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ των επιχειρήσεων. Γιατί πιστεύω ότι επιχειρήσεις μάλλον γιατί οι επιχειρήσεις είναι άρτα συνδεδεμένε με τις ρίζες μου, με τη ζωή μου. Και δεν πιστεύω ότι η κοινωνική καινοτομία έρχεται σε αντιπαράθεση με τις επιχειρήσεις, γιατί η κοινωνική καινοτομία δεν σημαίνει είμαι κοινωνικός, ε, έχω τάση δηλαδή προς την κοινωνική προσφορά μόνο, όχι. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι Μπορεί να φαίνεται σε αντιπαράθεση το ένα με το άλλο, αλλά η κοινωνική καινοτομία μετά από όλες τις μελέτες που έχω κάνει δεν είναι τίποτα άλλο από καινοτομία από κάτω προς τα πάνω. Είναι συμμετοχική καινοτομία. Οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την διαδικασία. Οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη διαδικασία, την προσέγγιση των χωρών μελών. Οι ερευνητές έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν την κατεύθυνση που θα πάρουν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει η καινοτομία. Οπότε είναι στοιχεία ενός συνόλου που μπορούν να βοηθήσουν το σύνολο αυτό να προχωρήσει και να πάει καλά και ακριβώς αυτό θέλουμε. Έτσι επανέρχομαι στο ρόλο του πολίτη που είναι πολύπλευρος. Πάντα για την κοινωνική καινοτομία. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Στα smart ε, τηλέφωνα υπάρχουν ε, διάφορες εφαρμογές και ποιος τις κάνει. Οι επιχειρήσεις, οι πολίτες, ακόμα και παιδιά. Και αυτό είναι η επιτυχία του iPad, των ε, έξυπνων τηλεφώνων, iPhone κλπ. Ότι δηλαδή οι ίδιοι πολίτες έχουν μια επιχειρηματική προσέγγιση. Αυτό είναι η κοινωνική καινοτομία. Είναι από κάτω προς τα πάνω, είναι συμμετοχική προσέγγιση όπου όλα τα στοιχεία της κοινωνίας συμμετέχουν. Αν βρούμε αυτή τη διατύπωση πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι. Οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όλοι θέλουμε την καινοτομία. Για μένα η καινοτομία τι είναι, είναι επιτυχία στην αγορά. Είναι μια νέα ιδέα η οποία επιτυχώς μπαίνει στην αγορά και χρησιμοποιείται στην κοινωνία. Συνεπώς, προσπαθώ να δείξω στην έκθεσή μου πόσο σημαντική είναι η επιχειρηματικότητα. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ επίσης για την καινοτόμο προσέγγισή σας στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε τελικά μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σκιώδη κύριε Σατόρη πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μέρκης για την εξαιρετική της δουλειά. Δύσκολη δουλειά και αυτή και των ε, άλλων εισηγητών. Εγώ συζήτησα με τους συναδέλφους μου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την έκθεση αυτή, έκθεση πρωτοβουλίας, προσπαθώντας να κάνουμε μια, να διανύσουμε μια απόσταση από τις αρχικές μας θέσεις και γι' αυτό καταθέσαμε και αρκετές τροπολογίες, πολλές από αυτές από κοινού. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας έχει την αξία θα έλεγα μιας εκθέσεως πλαισίου και γι' αυτό είναι περισσότερο μία έκθεση αρχών θα έλεγα και όχι τόσο μία έκθεση συγκεκριμένου περιεχομένου που να εδράζεται στην πραγματικότητα και τη συγκυρία. Γνωρίζει βέβαια η συγγήτρια ότι εμείς κάναμε μία προσπάθεια τις τελευταίες εβδομάδες όχι να αμφισβητήσουμε την κατεύθυνση που δίνει στην έκθεσή της, αλλά να προσπαθήσουμε να δούμε εάν θα ήταν χρήσιμότερο να συνοδεύσουμε τις εργασίες της Επιτροπής στον τομέα της λεγόμενης κοινωνικής καινοτομίας προτείνοντας την εκκίνηση ενός πιλωτικού προγράμματος το οποίο να ανοιχνεύει τις ορθές πρακτικές και τις χρήσιμες εμπειρίες στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν προσπαθήσουμε πριν προσπαθήσουμε λοιπόν να περάσουμε σε μία προσπάθεια με την οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι δηλαδή ο πολίτης είναι στο κέντρο των στόχων και της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και όταν μιλάμε για την παιδεία, τη γνώση, τα πανεπιστήμια, τον δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις. Πάντα στο κέντρο της ενασχόλησής μας είναι ο πολίτης αλλά πρέπει να προχωρήσουμε βέβαια γιατί βλέπουμε ποια είναι η αρμοδιότητά μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Εμείς εδώ βρισκόμαστε, το θυμίζω να μου το επιτρέψετε, όχι στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Δεύτερον, ο κοινωνικός τομέας αυτό που έχει ανάγκη είναι από πόρους. Έχει σημασία βέβαια να συμφωνούμε σε επίπεδο αρχών, αλλά θα πρέπει να ακολουθείται η συμφωνία αυτή από ένα ιστό θέσεων που να δίδουν εγγυήσει ε, για την κοινότητα των πολιτών που τη συναποτελούν. Βλέποντας λοιπόν τις προσδοκίες των πολιτών για μια πραγματική νέα βιομηχανική πολιτική, μια βιομηχανική πολιτική την οποία έχει ανάγκη σαν τον άρτο τον επιούσιο η Ήπειρος αυτή για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητη μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως το έχει προτείνει και η στρατηγική για την Ευρώπη του 20 και η στρατηγική για το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των φυσικών πόρων κτλ. Να περάσουμε λοιπόν μέσω της οικονομίας και μέσω ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού βιομηχανικού ιστού στις λεγόμενες καινοτόμες βιομηχανικές δραστηριότητες. Εδώ από τη μία εμείς συμμεριζόμεθα την ιδέα σύμφωνα με την οποία έχει σημασία να προωθήσει κανείς και το θέμα των κοινωνικών καινοτομιών, γιατί είναι καινοτομίε οι οποίες αφορούν την καθημερινότητά μας. Από την άλλη όμως πιστεύουμε το ότι να περιοριστούμε να πούμε μόνο αυτό, στην ουσία θα καταστήσουμε το θέμα της βιομηχανικής δραστηριότητας ένα από τα πάρα πολλά θέματα τα οποία, στα οποία στην συγκεκριμένη στιγμή η απάντηση και η κάλυψη των προσδοκιών της δεν είναι επαρκής. Γι' αυτό λοιπόν η κοινωνική καινοτομία από μόνη της, αν θέλουμε να επιβάλλουμε μόνο αυτό το θέμα προς συζήτηση, τότε φοβάμαι ότι παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα των τελευταίων ετών και αντίθετα θα ήθελα εγώ να βάλουμε σαν κεντρικό θέμα συζήτησης την βιομηχανική καινοτομία. Αυτή είναι λοιπόν μια πρόταση που κάνω και εγώ και οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες μας και ελπίζουμε έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συνενετική θέση και να συμβιβάσουμε ε, κάποιες θέσεις οι οποίες αυτές δεν είναι κακές αλλά είναι ελαφρά φιλοσοφικές. Σας ευχαριστώ. Μία σειρά συνάδελφων έχουν στήσει το λόγο. Στι είναι καταρθεί η Επίτροπο και θα έλεγα παρακαλώ ο καθένα δύο λεπτά. Ο κ. Τσουκαλά είναι ο πρώτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια μικρή παρατήρηση. Και η κυρία Σαρτόρη και η κυρία Μέρκης έχουν εστιαστεί στην έννοια του πολίτη. Το κέντρο όλων των προσπαθειών δεν είναι ο πολίτης, είναι ο άνθρωπος. Ο πολίτης είναι μια μικρή ιδιότητα της δημοκρατικής σου συγκρότησης. Δεύτερη παρατήρηση. Η καινοτομία αποτελεί πράγματι την απάντηση σε όλες τις μίζωνες κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντολογικές, επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κληθεί να απαντήσει και θα κληθεί να απαντήσει ακόμα εντονότερα και στο μέλλον. Παρόλα τα αυτά, εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η καινοτομία αποτελεί θεμελιώδη συνιστόσα του τριγώνου της γνώσης το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Η καινοτομία, όπως προσφυώς ελέγχθη, είναι η μετατροπή της γνώσης σε χρήμα, ενώ η γνώση και η έρευνα είναι η μετατροπή του χρήματος αυτές. Άρα το τρίγωνο αυτό έχει και την οικονομική διάσταση για όποιον έτσι θέλει να το ερμηνεύσει. Επομένως, η προσπάθειά μας πρέπει να είναι να ενισχύσουμε το τρίγωνο της γνώσης η Ευρώπη δεν είναι μια απομονωμένη νησίδα στον κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει να συγκρίνει τον εαυτό της και στην καινοτομική της διάθεση και στην ερευνητική της διάθεση με αυτά που σήμερα γίνονται στον κόσμο. Σε ποιον κόσμο, σε ένα κόσμο που έχει 7 εκατομμύρια επιστήμονες, που ξοδεύει ένα τρισεκατομμύριο το χρόνο για έρευνα και καινοτομία, έχοντας αυξήσει το ποσοστό από το 2002 κατά 45%. Έχουμε την άνοδο των ε, κρατών όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, κάθε μία από τις οποίες παράγει 1,5 εκατομμύριο επιστήμονες θετικών κατευθύνσεων και μηχανικούς το χρόνο, η Κίνα 2,5 εκατομμύρια και όπου το 20% των παγκόσμιων δημοσιευμάτων γίνεται από την Αμερική και το 50% από τις πατέντες κατοχυρώνονται ε, εκεί. Μία προσπάθεια του τύπου που προτείνει η κυρία Σαρτόρη στα πλαίσια του ανθρωπισμού της κυρίας Μέρκες θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη της αυτά τα στοιχεία που είναι όροι επιβίωσης για την Ευρώπη, για την καινοτομία και για τους στόχους της. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε. Danke, Kollege Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω να πω στην κυρία Μέρκης είναι ότι εξεπλάγει κάπως από το σχόλιο της που λέει ότι παρόλο που είναι στους σοσιαλιστές και δημοκράτες αγαπάει τις επιχειρήσεις. Κυρία Μέρκης, εσείς ως σοσιαλδημοκράτησα είσαστε υπερτροφοδότησης ενός κράτους που προσφέρει καλές υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία, ε, συντάξεις. Είσαστε υπέρ ενός τομέα που προστατεύει τον κόσμο και λαμβάνει υπόψη τα πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας μας. Για το σκοπό αυτό όμως το κράτος χρειάζεται πόρους και οι πόροι έρχονται από τους φόρους. Φόρους που πληρώνουν και οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι. Εσείς λοιπόν, σοσιαλδημοκράτησα, πρέπει να είσαστε υπέρ των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει απόλυτη συνοχή στο να είσαστε υπέρ των επιχειρήσεων ούσα σοσιαλδημοκράτησα. Πέρα τώρα από αυτή τη διευκρίνηση. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για την δουλειά που έκανε με τις 302 τροπολογίες που πήρε και από τις οποίες κατέληξε σε 35 συμβαστικές. Κάποιες από τις τροπολογίες μου συμπεριλαμβάνονται σε μερικές συμβαστικές. Θέλουμε να υπογραμμίζουμε το ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, ξέρουμε ότι η επιτυχία των μικρών επιχειρήσεων φαίνεται από την ε, οικονομική ανάπτυξη. Στόχος δηλαδή κάθε επιχείρησης μικρής είναι κάποια μέρα να γίνει μεσαία επιχείρηση και στόχος κάθε μεσαίας επιχείρησης είναι κάποια μέρα να γίνει μια μεγάλη επιχείρηση. Γι' αυτό και θέλω να δω τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ξεκίνησε πρόσφατα και που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τον Μάιο, ενώ το οποίο έχουμε και εμείς ψήφισμα. Η εισηγήτρια επίσης έχει συμπεριλάβει τι τροπολογίε μου που αναφέρονται στη σημασία των επενδύσεων, τη κατάρτιση των πολιτών, της χρήσης δηλαδή του ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτουμε, κάτι το οποίο αποτελεί κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Κυρίως επειδή η έκθεση αυτή έχει σαν στόχο να υπογραμμίσει τον ρόλο των πολιτών στην καινοτομία και να δείξει ότι ο καθένας έχει πρόσβαση στην καινοτομία και γεφυρώνεται έτσι η πορεία, η απόσταση ανάμεσα στην αρχική ιδέα και την εμπορία ενός προϊόντος. Και για την κυρία Σαρτο... με την κυρία Σαρτόρη συμφωνώ και με την κυρία Μέρκης που βλέπει πολύ βασικό στοιχείο της επιχειρήσης για την νέα στρατηγική μας για την ε, καινοτομία με τις παραγράφους 1, 7, 15, 19 και 22. Βασικό στοιχείο είναι η δημιουργία μιας επιχείρησης επίσης, πώς δημιουργείται. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, πιστεύω, και εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, η έκθεση αυτή θα πετύχει. Είναι στον σωστό δρόμο. Απ' την άλλη μεριά, στις παραγράφους 2, 4, 8 και 10 εξαπλάγει λίγο επειδή οι επιχειρήσεις και ο πολίτης μπαίνουν στο ίδιο Μάλλον το γεγονό ότι μπαίνουν στο ίδιο επίπεδο δεν έχει συμπεριληφθεί. Δεν έχουν συμπεριληφθεί δηλαδή στι συμβαστικέ αυτέ οι παράγραφοι. Εγώ το είπα και στην προηγούμενη συζήτηση ότι για μένα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ότι υπάρχουν κοινωνικέ επιπτώσει στην, από την καινοτομία. Και για να είμαστε συνεπείς με το προηγούμενο κείμενό μας, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιούμε την ιδέα της κοινωνίας της καινοτομίας γιατί συμπεριλαμβάνει και τον άνθρωπο και τις πνευματικές του ε, ικανότητες αλλά και τις δομές που έχουμε στις κοινωνίες μας επιχειρήσεις, σχολεία, συλλόγους ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι ο πολίτης μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες για να πετύχει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα προχωρήσουμε έτσι καλά με την εισηγήτρια και περιμένω να έχουμε την επόμενη συνάντηση σκιώδης με την εισηγήτρια. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της μας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέρκης για την έκθεσή της όσον αφορά τις κοινοτομίες και θα ήθελα να αναφερθώ στην σημασία της ε, τεχνολογίας ε, ενημέρωσης γιατί και το διαδίκτυο και το ευρυζωνικό φάσμα μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να βγει από την κρίση. Αυτά είναι μια πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας και μια που τα δίκτυα ενών υψηλή ταχύτητα είναι πάρα πολύ σημαντικά, μπορεί αυτά τα κανάλια να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη <clears throat> στο τομέα της ε, δημόσιας ε, διοίκησης, ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και η ηλεκτρονική εισφορά στον τομέα της δημόσιας υγείας. Και θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 7 της Κομισιόν, και τις τη κυρία Σαβέλη. Εμπνεόμενοι από αυτά που διαμήθησαν στις ΗΠΑ θα έλεγα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, γνώσει μα για να αξιολογήσουμε πολύ καλύτερα τη δυνατότητα χρήση των πόρων μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ να εξεταθούν καλύτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Στουσνόφσκι. E, e, Ευχαριστώ πρόεδρε. Σκιώδης συζητητής θα ήθελα να εγκομιάσω τις προσπάθειες της κυρίας Μέρκης ε, η οποία παρουσιάζει και τονίζει το τι είναι η καινοτομία. Αυτά είναι πάρα, πολύ σημαντικά για το μέλος της ε, Ευρώπης. Η δυνατότητα ανταγωνιστικότητας Ευρώπης εξαρτάται από την κοινωνία. Όπως και οι προλαλήσαντες, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Είναι περίπλοκο όταν θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της κοινωνικής καινοτομίας και να την αποχωρήσουμε από το σύνολο. Εμείς είμαστε υπέρ μιας πιο ευρείας ε, αντιμετώπισης της καινοτομίας και υποστήριξης της καινοτομίας. Οι καινοτομίες πάντα θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής και δεν θα πρέπει να τονίσουμε κάποια μορφή και να προτελήσουμε κάποια μορφή. σε επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, τονίζοντας ακριβώς τις κοινωνικές ε, πτυχές. Όπως είπαμε, οι μικρές επιχειρήσεις θέλουν να μεγαλώσουν, οι μεγάλες θέλουν να μείνουν ακόμα πιο μεγάλες. Το γεγονός ότι η κυρία Μέρκης τονίζει τις δραστηριότητες ε, κάποιων νέων φοιτητών στον τομέα του iPhone είναι κατά μας το πρώτο βήμα σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ πολύ αξιόλογο να ενισχυθούν οι κύκλοι καινοτομίας, να ενισχυθούν οι νέες ιδέες των πολιτών για να βελτιωθεί η ζωή. Έχω όμως ε, κάποιο πρόβλημα με το να τονίζεται τόσο πολύ η καινοτομία και η δραστηριότητα νομίζω από κάτω προς τα άνω είναι πολύ καλύτερος κινητήρας της αγοράς. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που οι συζητήσεις γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ πιο σοβαρό από ό,τι είχαμε φανταστεί στην αρχή. Γιατί όπως σας είπαμε καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η Ευρώπη και η θέση της στο μελλοντικό κόσμο εξαρτάται από αυτά και προτίθεμαι να συνεργαστώ ούτως ώστε η έκθεση να τονίσει ακόμα περισσότερο τη σημασία της καινοτομίας και θα ήθελα ευχαρίστως να υποστηρίξω στην κατεύθυνση αυτή την εισηγήτρια. η καινοτομία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Στη φάση αυτή που βρισκόμαστε εμφανίζονται διάφορα σημεία που είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα ότι η θεμελιώδης γνώση στην Ευρώπη πάει πολύ καλά, ενώ από την άλλη μεριά όταν περνάμε στην καινοτομία και στην εφαρμογή, εκεί μας χρειάζεται πολύς χρόνος συχνά και εκεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Δείτε και με την ευρυζωνικότητα για παράδειγμα ή στην υγεία ή για τους ηλικιωμένους. Υπάρχει κενό λοιπόν. Άρα, όντω αυτή η ένωση καινοτομία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Κάτι άλλο είναι ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που ακριβώς για την περίοδο 2014-2020 να φροντίσουμε να υπάρχει πρόγραμμα για την έρευνα και πόρη δηλαδή Όταν λοιπόν προταθούν αυτά, θα πρέπει να έχει προηγηθεί στην έκθεση κάτι πολύ συγκεκριμένο για αυτά, για να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει ζήτηση και για την κοινωνική καινοτομία. αλλά δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα πολλά πράγματα. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι αυτοί που είναι είτε βιομηχανία, είτε οι ίδιοι οι πολίτες που πρέπει να δούμε ότι καλύπτονται από το λεγόμενο διαμάντι. Εξού και δικές μου οι τροπολογίες που έχουν συμπεριληφθεί. Η έκθεσή σας είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγκαία, αλλά τουλάχιστον να μπορέσει να ερμηνευτεί στην πράξη με κάτι πιο συγκεκριμένο, οικονομικά δηλαδή, με οικονομικούς πόρους στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Ένα μικρό σχόλιο σχετικά με τον ορισμό της κοινωνικής καινοτομίας. Και οι δύο αυτές λέξεις χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο από αυτούς που τις χρησιμοποιούν. Πριν έρθω εδώ στο Κοινοβούλιο, πριν γίνω Ευρωβουλευτής, ήμουν πανεπιστημιακός γύρω από τέτοια θέματα ορισμών και είχα προσπαθήσει να ξεκαθαρίσω κάπως τα πράγματα γιατί υπήρχε μια σύγχυση σε επίπεδο ορολογίας. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι η κοινωνική καινοτομία είναι διαφορετική από την καινοτομία σε κοινωνικά θέματα. Η κοινωνική καινοτομία είναι καινοτόμες λύσεις σε ε, κατεπήγοντα κοινωνικά προβλήματα όπως η γύρανση του πληθυσμού χρησιμοποιώντας όμως περισσότερο το ισχυρό κοινωνικό ιστό και το κοινωνικό δίκτυ της κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών είναι ελαστική και ακριβώς ε, μια κοινωνία των πολιτών μη γραφειοκρατική μπορεί να συνεισφέρει καινοτόμες λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα. Δεν μιλάμε μόνο για καινοτόμε λοιπόν λύσει, αλλά και για τον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο οι λύσει αυτέ ε, επιβάλλονται. Βασίζονται σε κοινωνικά δίκτυα μέσα από τα οποία μπορεί κανείς ε, να συνεισφέρει την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό είναι ο ορισμό τον οποίο χρησιμοποιούν οι πανεπιστημιακοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στι ΣΥΠΑ, στι σκανδιναβικέ χώρε, και θα πρέπει νομίζω να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό όταν μιλάμε για κοινωνική καινοτομία και να μην έχουμε στο νου μας εντελώς διαφορετικά πράγματα. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τους όρους αυτούς έχω καταθέσει μια τροπολογία και νομίζω ότι η συγγήτρια την αποδέχεται σαν συμβιβαστική. Κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί έφτασα πολύ αργά, έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, ήμουν σε μία άλλη δυστυχώς συνάντηση. Δυστυχώς δεν μπορώ να παρευρίσκομαι σε δύο συνεδριάσεις ταυτόχρονα. Αλλά έχει μεγάλη σημασία η συγκεκριμένη έκθεση, γι' αυτό έπρεπε να είμαι εδώ έστω και τώρα. Η πρόταση της κυρίας Μέρκη είναι μια πρόταση περίπλοκη αλλά πηγαίνει προς την καλή κατεύθυνση σε σχέση με την καινοτομική Ευρώπη την οποία όλοι επιθυμούμε. Υποστηρίζω λοιπόν τις γενικές γραμμές της πρότασης. Υπάρχουν κάποιες επιμέρους διαφορές και γι' αυτό συζητάμε τις συμβιβαστικές προτάσεις. Πάντως συμφωνώ με την καινοτομία και στον κοινωνικό τομέα και την καινοτομία η οποία είναι ευεργετική για τον πολίτη. Ε, θα ήθελα επίσης να πω, όπως και η συνάδελφος Καρβάλιο, ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις ανάμεσα στην καινοτομία, στον κοινωνικό τομέα και στην κοινωνική καινοτομία. Η Καρβάλιο το είπε σωστά. Έχουμε να κάνουμε με μία έννοια πολύ ευρύτερη από την προηγούμενη που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα. Δεν θέλουμε μία πρόταση που να μην καλύπτει τις ανάγκες του μέλλοντος. ούτε θα πρέπει να φανούμε ιδιαίτερα περιοριστικοί στην παρουσίαση της έκθεσης και των τροπολογιών. Έχω την αίσθηση ότι οι βασικές γραμμές τις οποίες προτείνει η κυρία Μέρκης είναι αποδεκτές από πλευράς μας. Ναι λοιπόν στην κοινωνική καινοτομία, ναι σε μια καινοτομία η οποία να έχει σαν στόχο τον άνθρωπο, σαν έχει σαν στόχο, να έχει σαν στόχο τον πολίτη γιατί αυτό μας λείπει σήμερα τελικά. Και κάποια από τα κενά τα οποία έχουμε μπορεί να τα καλύψουμε αν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στους πολίτες. Υπάρχει αλλιώς ο κίνδυνος να κάνει κανείς κάποιες επιλογές οι οποίες ε, ε, να μην είναι ιδιαίτερα αποδοτικές στο μέλλον. Ελπίζω να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να επιλέξουμε καινοτομίε, οι οποίες να είναι διαρκείς. Ευχαριστώ. Στα σύνορα στην Κομισιόν, κύριο Στόρε, αν δεν κάνω λάθος. Thank you very much, Chairman. I know we are very short of time. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος περνάει. Θέλω να μεταφέρω ως μήνυμα ότι η Επιτροπή στηρίζει την έκθεση της ε, κυρίας Μέρκης και τις τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί. Κάποια σημεία τώρα που είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προϋποθέσεις πλαίσιο που αναφέρει και η κυρία Μέρκης, η πρόσβαση στα κεφάλαια, οι δημοσίες συμβάσεις, η διεθνής διάσταση, που τα είπε και ο κύριος Τσουκαλάς και η κυρία Μέρκης. Η κυρία Σαρτόρη τώρα και ο κύριος Βιντάλ Κουάρδας όταν ε, αναφέρθηκαν στις ε, τροπολογίες τους αναφέρθηκαν στην νομοθεσία για την καινοτομία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την Επιτροπή. Τώρα για τους ορισμούς δεν θα μπω στις ε, λεπτομέρειες, αλλά υπήρχε μια τροπολογία του κ. Χατζημαρκάκη, αν δεν απατώμε, που έλεγε ότι θα πρέπει να οριστεί από την Επιτροπή η, η καινοτομία. Έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να είναι πιο ρεαλιστική και να θέσει επιτάπητος, όπως προτείνουν διάφορες τροπολογίες, να θέσει επιτάπητος λοιπόν δίκτες. Ένα σύνολο δικτών που μας επιτρέπουν εμάς που παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις να μπορούμε να καθορίσουμε καλές πολιτικές για την καινοτομία. Εκεί που αναφέρεται τι κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο αυτό. Αυτό είναι κάτι που με απασχολεί πιο πολύ, γιατί δεν έχουν ζητηθεί εγγύσεις. Αυτό που έχουν ζητηθεί είναι δάνεια. Οι εγγύσει ίσως ε, επειδή υπάρχουν, δεν υπάρχουν δείγματα ότι βραχυπρόθεσμα θα ζητηθούν τέτοιες εγγύσει. Πάντως, στο νέο πλαίσιο ίσως υπάρξει κάποιο περιθώριο και για αυτές. Τέλος, για την καινοτομία και τα πανεπιστήμια και την επιχειρηματικότητα. Φυσικά και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπως λέτε και εσείς είναι πράγματα τα οποία μαζί πάνε. Είναι και αυτά ένα τρίγωνο, δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Είναι το διαμάντι όπως το είπε η ίδια συγκήτρια. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα η κυρία Βασιλείου Επιτρέπος μπορεί να σας πει πολύ περισσότερα για αυτά. Τελευταία ανησυχία εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει smart fiscal consolidation. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν ε, γίνονται περικοπές στον προϋπολογισμό για την έρευνα και την καινοτοπία και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσει τελικά. Αυτά ήταν τα σχόλια, αν δεν πατώ με τις κυρίες Σαρτόρη, που λέει ότι χρειάζεται σωστός προπολογισμό εφόσον θέλουμε ανάκαμψη. Σταματάω εδώ. Ευχαριστώ. Merci. Thank you very much. Ms. Merkes, once again. Η κυρία Ευχαριστώ συνάδελφοι για την εξαιρετική σας συνεισφορά στη συζήτηση. Η λογική σου θεωρείται επιτυχημένη μόνο στην περίπτωση που οι συνομιλητές σου μπορούν να εξηγήσουν ακριβώς αυτά τα οποία εσύ λες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσπάθεια την οποία κάνατε. Ευχαριστώ και συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Βέβαια μερικές φορές υπάρχουν κάποιες ιδεολογικές ε, μορφές περιορισμού αν θέλετε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες πιστώσεις. Νομίζω ότι δεν μας χωρίζει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, ιδιαίτερα σε μία πλευρά. Έχω την αίσθηση ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό συμφωνείτε με αυτά τα οποία προτείνω. Μιλάμε όλοι για την κοινωνική καινοτομία και υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία δεν αναφέρομαι και τα οποία μπορούμε όμως να μας βρουν σύμφωνος. Πράγματι η κοινωνική καινοτομία είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που δημιουργούνται στον κοινωνικό τομέα. Δεν μιλάμε κοινωνικά θέματα ή τις κοινωνικές συνέπειες, αλλά προσπαθούμε να συμμετέχουμε σαν ομάδα στα πλαίσια μιας διαδικασίας που εξελίσσεται. Είναι δύσκολο να ορίσει κανείς τι είναι η κοινωνική καινοτομία και είναι επίσης δύσκολο να δώσει μια διαφορετική ονομασία. Ας μην προωθούμε λοιπόν, όπως είπε ο κ. μία μορφή καινοτομία εις βάρος άλλης, γιατί χρειαζόμαστε όλες τις μορφές καινοτομίας που υπάρχουν και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μια τροπολογία η οποία δείχνει ότι χρειαζόμαστε όλα αυτά τα στοιχεία για να είμαστε επιτυχείς. Εκεί βρίσκεται η ισορροπία θα έλεγα της καινοτομίας, πρέπει να διασφαλιστεί η ισορροπία αυτή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με επιτυχία στην αγορά. Υποστηρίζω λοιπόν την γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρειάζεται μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική. Συμφωνώ μαζί σας ε, κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής και συμφωνώ επίσης με τις διαδικασίες flagship για τη βιομηχανική πολιτική διότι θα έλεγα ότι συμβαδίζουν αυτά τα δύο, αυτές οι δύο διαδικασίες και θα μας διασφαλίσουν μια σωστή παρουσία της βιομηχανίας όχι σαν μία από τις πλευρές αλλά την καθοριστική. Σας ευχαριστώ που το υπογραμμίσατε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσουκαλά σχετικά με την ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης σχετικά με τη λεγόμενη ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων χρειάζεται αυτό για να καλύψουμε όλα τα κενά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Και αν έχουμε αφήσει έξω τα θέματα της ευφυούς ε, fiscal consolidation τότε ίσως είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε συμφωνήσει απόλυτα, εφόσον συμφωνήσουμε όμως θα τη συμπεριλάβω. Θα ήθελα να σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστήσω κυρία Μέρκες. Ιδίω και επειδή προσφέρεστε να βρείτε ευφυεί λύση για πιο δύσκολα ακόμα θέματα, μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ την εξέταση αυτού του σημείου τη ημερησία διάταξη. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε στι 12 Απριλίου μια επιτυχή ελπίζω έκταση και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέσα της διάταξης και να καλωσορίσουμε εγκαρδιότητα την Επίτροπο κυρία Βασιλείου δεν έρχεται συχνά σε εμά όπως άλλοι επίτροποι λόγω των θεμάτων βέβαια που μας απασχολούν υπάρχει όμως ένα θέμα για το οποίο μπορούμε πολύ καλά να συνεργαστούμε γιατί σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Δεν θέλω να το αναπτύξω. Σα χαιρετίζω. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Επιτροπή, που σα δω και θα ήθελα να σα δώσω το λόγο για κάποια εισαγωγικά σχόλια. Παρακαλώ. Ε, uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να σας μιλήσω για κάτι το οποίο με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος και που είναι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το λεγόμενο EIT. Είναι ένα από τα σχέδια τα οποία μας βοηθούν να φτιάξουμε το μέλλον μας. Γιατί μπορεί να κάνει τη διαφορά όσον αφορά το τοπίο το ευρωπαϊκό καινοτομία και να ενισχύσει την καινοτομία στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομία και Τεχνολογία δείχνει πώς εμείς οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της καινοτομίας ενωμένη προς έναν κοινό στόχο, αλλά και με ελαστικότητα για να σεβαστούμε την ποικιλομορφία των διαφόρων φορέων. Τα τελευταία χρόνια το Ίδρυμα αυτό ξεκίνησε από μια ιδέα και έγινε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Ξέρω ότι ορισμένοι από εσά στην Επιτροπή αυτή συμμετείχατε ιδιαίτερα δραστήρια προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο Καινοτομία και Τεχνολογία και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Σήμερα το Ίδρυμα αυτό μπορεί να εξακολουθεί να είναι ένα μικρό, αλλά μεγαλώνει συνέχεια. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να το τροφοδοτούμε, να το φροντίζουμε και σίγουρα θα μπορέσουμε να υποφεληθούμε και από τους καρπούς του σύντομα. Έχουμε μια καινοτόμα κοινωνία. Έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Αυτού Ιδρύματος και εργαζόμενους που με καινοτομία δουλεύουν σε τρεις τομείς που είναι τα λεγόμενα KICS, δηλαδή κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, οι οποίες βοηθούν οι διάφορες πλευρές να συμμετέχουν, να συνεργάζονται για την εκπαίδευση, για την ενέργεια και την έρευνα σε τομείς που είναι ζωτική σημασία για το κοινό μας μέλλον. Έτσι λοιπόν έχουμε τρία κικς όπως σας είπα. Το ένα είναι για την βιώσιμη ενέργεια. Το λεγόμενο κικ είναι energy. Το δεύτερο αφορά τις κλιματικές αλλαγές, το climate kick. Και το τρίτο είναι η μελλοντική κοινωνία πληροφόρησης και επικοινωνίας που ονομάζεται EIT ICT Labs. Μέσα σε 10 μήνες, χρόνο ρεκόρ πιστεύω, για κάτι τόσο περίπλοκο, τέτοιες εταιρικέ ε, σχέσεις τόσο περίπλοκες, έχει προχωρήσει, έχουν ξεκινήσει ήδη τα κίξ αυτά και έτσι έχουμε φτιάξει ένα μοναδικό ευρωπαϊκό μοντέλο αλληλοεπίδρασης μεταξύ των ε, φορέων του τριγώνου της γνώσης. Πρώτα απ' όλα τα ΚΙΚΣ θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις με την πρόθεση μιας νοτροπίας επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, το ΚΙΚ για την βιώσιμη ενέργεια, το ΚΙΚ in Energy, φροντίζει για 20 startup και spin-ups για την περίοδο 2011 με 2013. Τα διάφορα kicks αποτελούν κίνητρο για να ακολουθήσουν τη λογική μας οι επιχειρήσεις. Αποτελούν ε, ξεχωριστές νομικές ε, οντότητες με δική τους διάρθρωση και με πλήρη απασχόληση ε, διευθυντές. Η συνεργασία είναι χαλαρή. Θέλουμε εδώ να προσελκύσουμε την επιχειρηματική κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει κατά 25% στο συνολικό προϋπολογισμό των ΚΙΚΣ, κάτι που αποτελεί σημαντικό κίνητρο για να βρούνε από άλλες πηγές χρήματα, επενδυτές κλπ. Δεύτερον, τα ΚΙΚΣ δεν αποτελούν εικονικά μόνο δίκτυα, διότι γεωγραφικά έχουν μια συγκεκριμένη βάση διότι βρίσκονται σε τοπικές κοινότητες και το κάθε ΚΙΚ έχει 5 με 6 κέντρα με τα οποία συνεργάζεται όπου συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, ερευνητικά κέντρα αλλά και επιχειρήσεις και συνεργάζονται πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο ΚΙΚ. Με τα τρία αυτά ΚΙΚ έχουμε 16 τέτοια κέντρα από την Βαρκελόνη μέχρι το Βερολίνο και από την Στοκόλμη μέχρι τη Σιλεσία. Έτσι δημιουργούνται ομάδες καινοτομίας, clusters. Τρίτον, εκπαίδευση. Αυτή είναι η καινοτομία βασικά της ιδέας. Η εκπαίδευση συχνά είναι αυτό που λείπει σε πιο κλασικού τύπου εταιρικές σχέσεις. Με τα όμως και για πρώτη φορά εμείς προτείνουμε το τρίγωνο αυτό της γνώσης να συμπεριλαμβάνει εξίσου και τα τρία, και την έρευνα δηλαδή και την καινοτομία και την ανώτατη εκπαίδευση στον ίδιο βαθμό. Τα ΚΙΚΣ έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα με ε, ακαδημαϊκούς και πανεπιστήμια. Υπάρχουν μαθήματα masters, υπάρχουν ε, μετεπτυχιακά, υπάρχουν summer schools θερινά πανεπιστήμια. Το ΚΙΚ για την ενέργεια, για παράδειγμα, με την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει 2.000 φοιτητές για τα επόμενα τρία χρόνια. Το συγκεκριμένο αυτό ΚΙΚ λοιπόν για τη βιώσιμη ενέργεια θα ξεκινήσει το φθινόπωρο με τα προγράμματα Masters και τα άλλα δύο θα ακολουθήσουν του χρόνου. Αυτά τα νέα προγράμματα επικεντρώνονται στις ε, τεχνολογικές ικανότητες αλλά και στην επιχειρητικότητα ή την ε, επιχειρηματική ανάπτυξη και ενισχύουν την κινητικότητα των εταίρων μεταξύ των διάφορων ΚΙΚ σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις ή σε εταιρικέ σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι Υπάρχει μια διάδραση μεταξύ των διαφόρων ε, τομέων που ανταποκρίνεται στη ζήτηση από την αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί αν θέλουμε να αλλάξει καινοτροπία των ε, νέων μας και να ανταμείψουμε την επιχειρηματικότητα. Πέρα όμως από τα ΚΙΚΣ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας είναι και ένας ζωντανό οργανισμός. Οι υπηρεσίες του ε, δρεύουν στην Βουδαπέστη εδώ και ένα χρόνο και λειτουργούν εκεί. Οι προσλήψεις συνεχίζονται και στα τέλη της χρονιάς το Ινστιτούτο αυτό θα έχει φτάσει σε ένα σημείο που θα λειτουργεί πια κανονικά. Τέλος, το Ίδρυμα, το Foundation για το EIT έχει ξεκινάσει τις εργασίες του έτσι όπως προβλέπεται στον σχετικό κανονισμό. Το Foundation αυτό, το Ίδρυμα, είναι άλλο ένα στοιχείο καινοτόμο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Καινοτομία και την Τεχνολογία θα βοηθήσει και τα ΚΙΚΣ να προσελκύσουν πόρους από τον ιδιωτικό τομέα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορώ να πω ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται από πολύ έμπειρες προσωπικότητες υπό την ηγεσία του Προέδρου του κυρίου Κρίστιαν Ζουργένα που είναι και διευθυντής της ΟΛΒΕ. Κυρίες και κύριοι, είπα στην αρχή ότι προχωράει και μεγαλώνει ότι σε μας έγκυται πια να το κάνουμε να ανθίσει. Και όπως είπε και ένας εδώ στην Επιτροπή σας πρόσφατα, η κυρία Καλβάλιο, επιτρέψτε μου, όπως το είπε, είπε αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή σε εμά επόκειται να το αφήσουμε να ενθύσει. Τώρα θα περάσω σε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, για το Δεκέμβριο. Θα υποβάλω σε εσά την πρώτη στρατηγική καινοτομία, την ατζέντα δηλαδή για τη στρατηγική καινοτομία που θα αναφέρει τις προτεραιότητές μας για τα επόμενα 7 χρόνια. Θα επικεντρωθούμε σε διάφορα θέματα για τα ΚΙΚΣ, όπως επίσης και στις ε, στρατηγικές δραστηριότητες που θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να υποβάλω πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Καινοτομίας και Τεχνολογίας εκεί που χρειάζεται. Φυσικά και θα βασιστώ στις εμπειρίες που είχαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των ΚΙΚΣ και έτσι θα φροντίσουν να εφαρμοστούν και να γίνουν αλλαγές ώστε να λειτουργήσει αυτό ακόμα πιο αποτελεσματικά. Βασίζομαι στη στήριξη της δικιάς σας Επιτροπής στο εγχείρημα αυτό ώστε να μπορέσουμε μαζί να δώσουμε την νέα μορφή στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογία. Επίσης, η χρονιά αυτή είναι αποφασιστική σημασίας για το τι τύχη περιμένει το ΙΑΕΤ e στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ελπίζω ότι, όπως λέει και η Επίτροπος, η συνάδελφός μου και ο Γκαν Κουίν, θα προχωρήσουμε σε συνεργασία και θα έχουμε ένα κοινό σκοπό. Ελπίζω να μπορέσουν να υπάρξουν συνέργειες και να έχουμε ένα πεδίο καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη συνοχή. Ελπίζω ότι θα έχουμε στενή, στενή συνεργασία και με άλλους παράγοντες. Στηρίζω απόλυτα την προσέγγιση αυτή. Όμως πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι για την προσθεθέμενη αξία που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα καινοτομία και Τεχνολογίας στο πεδίο αυτό ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνης. Το Ίδρυμα αυτό μπορεί να επηρεάσει μόνο εφόσον παραμείνει ελαστικό, ευέλικτο, που δεν θα περιοριστεί από τον κλασικό δρόμο χρηματοδότησης. Μην ξεχνάμε ότι έχει μια προσέγγιση που προσανατολίζεται περισσότερο στην επιχειρηματικότητα και στα αποτελέσματα. Τα ΚΙΚ συνδέονται άμεσα με τον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται λοιπόν μια ευελιξία στη δομή του, στη διακυβέρνησή του και στην λειτουργία του, αλλά και στην χρηματοδότησή του. Δεν θέλουμε επιπλέον βάρος εμείς στα ΚΙΚΣ που θα τα κάνει λιγότερο ελκυστικά και θα αντιβαίνει στον ίδιο τον στόχο και τον σκοπό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Καινοτομίας και Τεχνολογίας γι' αυτό και συνεργάζομαι στενά με την Επίτροπο Γκέργεν Κουίν. Είμαι πεπισμένη επίσης ότι μπορώ να βασιστώ στην πραγματογνωμοσύνη τη δικιά σας, των μελών της Επιτροπής αυτής, για να βρούμε έναν ευφύ τρόπο να χρηματοδοτήσουμε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας με ελαστικότητα και αυτονομία, πράγματα που είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία του. Τώρα μπαίνουμε σε ένα αποφασιστική σημασία σε στάδιο όσον αφορά το μέλλον του. Όπως ε, έχω πει και στους διευθές των ΚΙΚΣ, που τους είδα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα που τέλειωσε η περίοδος του setup, Τώρα πρέπει να αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα. Βασίζομαι στην συνεργασία μαζί σας και στην πολιτική στήριξη προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Καινοτομία Τεχνολογίας και το μέλλον της στρατηγικής του και της χρηματοδότησής του επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ και εισαγωγικά μπορώ να σας πω ότι η δική μας Επιτροπή ε, πάντα πραγματικά παρακολουθούσε την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Οικονομία και Τεχνολογία. Ορισμένοι από εμά μάλιστα είχαν τη δυνατότητα επιτόπου στη Βουδαπέστη να το επισκεφθούν και είμαι σίγουρο ότι αυτό είναι ένα σχέδιο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, η συνάδελφοι θα έχω το λόγο. Συνάδελφο Μπύρη, πρώτο. Έξι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ να υποβάλλετε σύντομε και εφής ερωτήσεις για να μπορέσει να απαντήσει μετά η Επίτροπο. Ναι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω καρδιότατα την Επίτροπε. Εγώ δεν έχω ερώτηση, μια παράκληση όσον αφορά την έναρξη εργασία του ε για τα ΚΑΠΑΤΑΦ. Και θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή κάτι άλλο που να μπορέσει να παρουσιαστεί στο δικό μας επαγγελματικό σύστημα, ούτως ώστε οι καθηγητές και οι φοιτητές να μπορέσουν γλίγορα να ωφεληθούν από τις νέες αυτές γνώσεις που απορρέουν. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποια πολιτική ούτω ώστε οι γνώσει αυτές να προωθούν σε εκείνου που θα μπορούν να ωφεληθούν από αυτέ. Αυτό θα ήταν νομίζω μια τεράστια πρόκληση και για τον τομέα τη παιδεία. Ευχαριστώ. Ο κ. Τσουκαλά έχει το λόγο. Να καλωσορίσω και εγώ κύριε Πρόεδρε την κυρία Επίτροπο. Είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι η Επίτροπος για την εκπαίδευση, στον πολιτισμό, την πολυγλωσία και την νεολαία φαίνεται να είναι ταυτοχρόνως υπεύθυνη και για το EIIT, το οποίο εγώ το είχα καταλάβει να είναι ένα καινοτομικό και ερευνητικό κέντρο το είχα παρακολουθήσει όταν συνίστατο υπό την προεδρία του κυρίου ε, ε, Φώτη Καφάτου, του πρώτου πρόεδρου. Ε, και τώρα μια απλή ερώτηση. Ξανά ότι θεωρώ πολύ, πολύ καλό προχώρημα όχι τη σύνδεσή του με την εκπαίδευση, αλλά τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό. Τα προβλήματα όμως που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη είναι τα προβλήματα να συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο καταμερισμό της καινοτομίας και της έρευνας. Αυτό η Ευρώπη παρά τις διακηρύξεις της, εγώ επιμένω να λέω ότι δεν το έχουμε πετύχει. Τα νούμερα παραδείγματι γιορτάζουμε για το EIT, αλλά εγώ να σας θυμίσω ότι ο Ομπάμα ίδρυσε 70 EIT στην Αμερική και ότι η Ινδία έχει 12 τέτοια, ότι οι δημοσιεύσεις, οι ερευνητικές της Κίνας για πρώτη φορά υπερέβησαν των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι πατέντες εξακολουθούν να κατοχυρώνονται 50% στην Αμερική. Θα ήθελα λοιπόν, μια που έχω εδώ την κυρία Βασιλείου, να μας πει εάν η συντονισμένη πρακτική που έχουμε τώρα για το 2020, λέμε το όραμα του 2020 διαδέχτηκε το θνησιγενές στη στρατηγική της Λισαβόνας του 2010. Θα αυξήσουμε την ένταση της προσπάθειας. Θα μπορέσει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί πράγματι. Αυτή είναι η κύρια και τελική μου ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Ξέρω ότι λειτουργεί ω ε, σώμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι εσεί το εφαρμόζετε αυτό πάρα πολύ. Έχω μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Παρατήρηση. Πράγματι η Επιτροπή αυτή βρίσκεται στο δύσκολο στάδιο, θα έλεγα, όπου υποστηρίζει. Υποστηρίζει την πτυχή της καινοτομίας μέσω τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή των ΚΙΚΣ. Ρωτάω τώρα, όπως λέει και ο κύριος Τσουκαλάς, όντως υπάρχει πολλή κίνηση στο δρόμο, σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε εξελίξεις πάρα πολύ γρήγορες, έχουμε κέντρα αριστείας, και πρέπει και εμείς να βρούμε τη θέση μας. Η Επίτροπος λέει ότι θέλουμε να έχουμε τις δικές μας δραστηριότητες, τις δικές μας ρυθμίσεις. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι σε όλο αυτό το φάσμα ευρωπαϊκών ε, μέσων που έχουμε, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, τις διάφορες ε, κοινέ πρωτοβουλίες, πλατφόρμες κτλ. Καταλήγουμε σε κάποιες επικαλύψεις και δεν είμαστε πιο ευάλωτοι. Ναι μαζί, αλλά όχι με επικαλύψεις. Υπάρχουν ένα σωρό παρόμοιες πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είμαστε πιο ευάλωτοι. Η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ, Επίτροπε που είστε μαζί μας και είναι σύμπτωση που έρχεστε την ίδια στιγμή που συζητήσαμε και το θέμα της καινοτομίας στην Ένωση. Η ερώτησή μου είναι η εξής λοιπόν. Πώς στα πλαίσια της αντίληψής σας το EIT ευθυγραμμίζεται με τις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ένωση για την Καινοτομία. Η Ένωση για την Καινοτομία αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά θέματα, προκλήσεις και το έχουμε συζητήσει αυτό στην έκθεσή μου. Τα EIPs, οι εταιρικέ αυτές σχέσεις, είναι εκεί για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία αν αγνοήσουμε τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, τότε θα πρέπει να στοχεύσουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Το θέμα της τεχνολογίας, σαν παράδειγμα, και της πρόσβασης στην τεχνολογία. Πώς λοιπόν τα ΚΙΚΣ μπορεί να ευθυγραμμιστούν με το EIPs. Μπορεί να είναι τμήμα των EIPs, κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να είναι χρήσιμο και το πώς θα τοποθετήσει κανείς τα EIT για, στο πολιετές πλαίσιο. Τι σημαίνει αυτό το οποίο είπατε για το πολιετές πλαίσιο. Πράγματι η καινοτομία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει κανείς εκ των προτέρων και όσο πιο ευέλικτος είναι κανείς τόσο πιο ε, περισσότερο επιταχύνει τις ε, καινοτομικές εξελίξεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, ευέλικτα μέσα για να προχωρήσουμε. Τα EIT μέχρι τώρα δεν έχουν επιδείξει την απαιτούμενη ευελιξία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προωθήσει κανείς αυτή τη νέα ιδέα σε κάποιες ε, μορφές κίνησης. Αλλά πάντως, έστω και με τον νόμο της βαρύτητας, ε, η δυσκολότερη στιγμή είναι η στιγμή της εκκίνησης, πριν αποκτήσει η διαδικασία κάποια ταχύτητα αφεαυτής. Μπορείτε λοιπόν εμείς να μας πείτε πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την ευελιξία την οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε. Hvala σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας ε, επίτροπε, ήμουν σκιώδης εισηγήτρια στο συγκεκριμένο θέμα από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Νομίζω ότι οι προτάσεις για το Ινστιτούτο μπορεί να συγκεκριμενοποιηθούν με σωστό τρόπο. Έχω πέντε ερωτήσεις να σας θέσω. Εσείς αναφερθήκατε, Επίτροπε, στο στρατηγικό ε, πρόγραμμα έρευνας. Υπάρχουν προγράμματα έρευνας τα οποία είναι σχεδιασμένα μέχρι το 2020 έχουν συμπεριληφθεί επίσης και προτάσεις στο roadmap με στον οδικό χάρτη μέχρι το 2050 με τα kicks τώρα. Τι γίνεται. Ε, ποια είναι η αντίληψη που έχετε για τα kicks. Πώς θα συνδέσετε τα EIT, παράδειγμα, με τη δική μας στρατηγική αντίληψη μέχρι το 2020 και μετά. Άλλο θέμα σχετικά με το Ινστιτούτο ε, προτείνονται κάποιες αλλαγές. Τι θέλετε ακριβώς να τροποποιήσετε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες εξηγήσεις. Τρίτη ερώτηση. Υπάρχουν 16 τέτοια κέντρα, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια του λεγόμενου Ινστιτούτου. Μπορείτε να μας ε, ε, μιλήσετε λίγο για τη γεωγραφική κατανομή των 16 αυτών κέντρων όπως επίσης και ποια είναι η λεγόμενη θεσμική κατανομή των δραστηριοτήτων. Πώς οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων αυτών κέντρων εντάσσονται και ενσωματώνονται στις, στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα κτλ. Μια επιπλέον ερώτηση. Στο, παρόν νομοθετικό πλαίσιο μιλήσατε επίσης και για τις ετικέτες EIT. οι οποίες θα πρέπει να εισαχθούν σε μια πρώτη φάση, σε εθελοντική βάση. Τι ακριβώς ε, σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με αυτό και κατά πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει την έρευνα. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μια ερώτηση. Νομίζω κύριε Επίτροπε ότι το EIT είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σχέδια που έχουμε. Έχετε κάποια ιδέα όσον αφορά την χρηματοδοτική πλευρά. Όχι να μας αναφέρετε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αλλά λίγο πολύ υπάρχει κάποια χρηματοδότηση για την επόμενη περίοδο, γιατί και βάσει αυτό θα αποφασίσουμε αν θα δώσουμε κάποια σειρά προτεραιότητας μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ε, καινοτομίας και έρευνας. Τελευταία κυρία Καβάλιο. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο που είναι ανάμεσά μας σήμερα. Καταρχά να ζητώ συγγνώμη αλλά έπρεπε να πάω στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. So I had to be there. Uh, but I just want very briefly uh, to... Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Επίτροπο Βασιλείου ε, EIT is ε, σε σχέση με τα EIT. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και βρισκόμαστε στην πρώτη φάση βέβαια, αλλά αυτή η πρώτη φάση είναι ταυτόχρονα και μια κρίσιμη φάση. Γιατί ε, νομίζω ότι μπορούν να αναπτυχθούν σωστά. Έχουμε μπροστά μας στο Κοινοβούλιο κάποιες συγκεκριμένες προκλήσεις, έχουμε την στρατηγική, έχουμε ε, κάποιες πρώτες δημοσιονομικές καλύψεις, ε, τον προϋπολογισμό δηλαδή. Συνεπώς βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση και μπορούμε νομίζω σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αρμόδια να ενισχύσουμε τη διαδικασία αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια για τις προτάσεις τις οποίες έκανε σχετικά με τη δημιουργία της ομάδας φίλων του EIT και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί έτσι μια ομάδα η οποία θα διευκολύνει τις συζητήσεις σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους συναδέλφους και θα υπάρξουν προτάσεις χρήσιμες ιδιαίτερα για το θέμα της χρηματοδότησης. Ήδη στην έκθεση Γαρίγα Πολέντο υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την χρηματοδότηση του EIT από τους προϋπολογισμούς μετά το 2013. Λοιπόν, η βασική ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη αυτού του μέσου και να συνεισφέρουμε έτσι στην καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας συνδράμουμε όσο μπορούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε πάρα πολλές προτάσεις, πολλές παρατηρήσεις, πολλές ιδέες. Νομίζω ότι η Επίτροπος τώρα καλείται να ανταποκριθεί και να απαντήσει κάποια από τα θέματα αυτά. θα ήθελα να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω που δεχθήκατε να προεδρεύσετε της ομάδα των φίλων του EIT. Η ομάδα αυτή είναι ανοιχτή σε όποιον ενδιαφέρεται και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερα σχετικά με το EIT και να το βοηθήσει. Έχει γίνει μέχρι συνάντηση εδώ και λίγες εβδομάδες. Προγραμματίζουμε μια δεύτερη συνάντηση γύρω στα τέλη του μηνός Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής σκοπεύω να προσκαλέσω ε, τους ε, υπεύθυνους διευθυντές των τριών ΚΙΚΣ έτσι ώστε να έρθουν να συναντηθούν με τα μέλη της ομάδας των φίλων, των EITs και να γίνουν κάποιες συζητήσεις για το πού βρισκόμαστε και τι πρόοδος έχει υπάρξει. Έχει σημασία λοιπόν να υπάρξει επικοινωνία με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα ΚΙΚΣ. Θα σας ενημερώσω το ταχύτερο δυνατόν ε, για τις ε, ημερομηνίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση για τις παράλληλες ή ανάμεσα στις παράλληλες πρωτοβουλίες οι οποίες εξελίσσονται όπως επίσης και στον διαφορετικό χαρακτήρα τον οποίο παρουσιάζει το EITs. Για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνουμε την παιδεία, την ανώτατη παιδεία, σε αυτή την εταιρική σχέση. Νομίζω ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για την επίτευξη των στόχων που περιλαμβάνει η στρατηγική μας για το 2020. Η παιδεία όπως γνωρίζετε είναι στην καρδιά αυτής της στρατηγικής. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να πιέσουμε θα έλεγα προς την χρήση των βέλτιστων μέσων. Καλά ότι φυσικά και υστερούμε στην Ευρώπη κατά πολύ στο ε, θέμα της καινοτομίας και της έρευνας ε, αλλά ακριβώ αυτός είναι ένας τρόπος για να δώσουμε έμφαση. Και όταν καλούμε τώρα τις κυβερνήσεις να κάνουν οικονομίες στι διάφορα, του ε, στις εθνικές τους οικονομίες. Τρεις τομείς τους ενθαρρύνουμε να επενδύσουν περισσότερα. Και αυτοί οι τομείς είναι ο τομέας της καινοτομίας, ο, και, ο τομέας της έρευνας και ο τομέας της, ε, της Και φυσικά παιδεία είναι σε όλα τα επίπεδα, αλλά σε αυτήν τη συγκεκριμένη προσπάθεια του EIT είναι, μιλούμε για ανώτερα εκπαιδευτικά συστήματα. Ε, Θα ήθελα να αποκλίνω λίγο από την άποψη της κυρίας Μέρκης γύρω από τις ε, κοινωνικές προκλήσεις. Έχω την αίσθηση ότι τα τρία κικς προσπαθούν να καλύψουν ε, κάποιες πολύ σημαντικές ε, κοινωνικές προκλήσεις. Η ενέργεια, ιδιαίτερα μετά από τα τελευταία γεγονότα στην Ιαπωνία, έχει καταστεί ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα, η κλιματολογική αλλαγή επίσης. Και πιστεύουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα που έχουμε για τον τομέα της παιδείας μας στον συγκεκριμένο χώρο είναι, είναι τα ICT. Και ακριβώς θα ζητήσω το ΚΙΚΑ ICT να με βοηθήσει έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν την εκπαίδευση ICT ε, στην, ε, στα επίσημα προγράμματά τους. Έχει σημασία να δώσουμε την όθηση αυτή στα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Σχετικά με το μέλλον, νομίζω ότι η Διευθυντική Επιτροπή του EIT θα κάνει προτάσεις για τους τομείς τους οποίους θα ήθελαν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους. Αυτές τις προτάσεις θα τις παρουσιάσουμε τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δει από εκεί και πέρα για το ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι έγκυρες και ποιες από τις προτάσεις αυτές καλύπτουν ε, τις κοινωνικές προκλήσεις γιατί εκεί βρίσκεται ένας βασικός στόχος του EIT. Και φυσικά όταν παρουσιάσουμε τις στρατηγικές μας σε εσά και στο Συμβούλιο θα πρέπει και εσείς να τις συζητήσετε. Μαζί μας ελπίζω. Εν τω μεταξύ θα υπάρξει μία περίοδος διαβούλευσης τέλος Μαΐου αρχές Ιουνίου θα είστε προσκεκλημένοι και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά με το μέλλον στον συγκεκριμένο χώρο προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα πρέπει να αυξήσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τα μελλοντικά kicks. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν άλλα 10 kicks ας πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε αργά αλλά σταθερά ναι με να υπάρξουν ορισμένα επιπλέον kicks αλλά όχι πάρα πολλά για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε και να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σχετικά τώρα με το τι προτάσεις ε, ε, θα κάνω. Αυτό θα εξαρτηθεί αν πολλής από την αξιολόγηση την οποία κάνουμε σε αυτή τη φάση. Ήδη έχουμε ζητήσει από εμπειρογνώμονες να μας πούν πώς έχουν αναπτυχθεί τα ΚΙΚΣ, Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΚΙΚΣ και πώς μπορούμε να αλλάξουμε κάποια θέματα τα οποία θα διευκολύνουν την μελλοντική ανάπτυξη των ΚΙΚΣ. Σχετικά με τις συνεργασίες, έχω κάποια κείμενα εδώ τα οποία σας δίνουν τις βασικές πληροφορίες των τριών ΚΙΚΣ. Ε, ποια είναι τα όργανα που συνεργάζονται μαζί τους κτλ. Θα σας τα αφήσω και μπορείτε να τα διανύμετε η γραμματεία σας στα μέλη της Επιτροπής σας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πω πάντως, ότι σε κάθε περιοχή όπου υπάρχει ακριβώς μια τέτοια συνεργασία, υπάρχει μια πολύ στενή επαφή ανάμεσα στα ιδρύματα ε, ανώτατης εκπαίδευσης, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα της συγκεκριμένης περιοχής. Θέλουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε το τρίγωνο γνώσης στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών και όπως σας είπα υπάρχουν 16 τέτοια σημεία στον ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο. Η ετικέτα EIT όπως είπατε πάρα πολύ σωστά εκδίδεται σε αυτή τη φάση σε εθελοντική βάση. Αλλά πολλά πανεπιστήμια έχουν υιοθετήσει την ιδέα και αυτά τα οποία είναι διατεθειμένα να ξεκινήσουν με το Ευρωπαϊκό Μάστερ θα βάλουν τη συγκεκριμένη ετικέτα, τον συγκεκριμένο τίτλο. Νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Χρειάστηκαν 10 μήνες για να καταλήξουμε στην υπογραφή της συμφωνίας και για να δοθούν οι πρώτες υποτροφίες, αλλά κάθε αρχή και δύσκολη. Ιδιαίτερα όταν έχει να ασχοληθεί κανείς με κάτι το τόσο καινοτόμο θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε είναι καινοτόμο, αλλά ταυτόχρονα είναι και φιλόδοξο και ελπίζω στο μέλλον να διαπρέψει. Από τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας και από τον τρόπο ε, πορείας μέχρι τώρα, από την πορεία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα, έχω εμπιστοσύνη στο μέλλον. Ελπίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας. Σχετικά με το θέμα της χρηματοδότησης συμπληρώνω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι κάτι το οποίο είπα και πριν. Εμείς δίνουμε το 25% της χρηματοδότησης, αλλά αυτά είναι χρήματα τα οποία επιτρέπουν την από εκεί και πέρα <clears throat> μόχλευση έτσι ώστε να προσελκυστούν πιστώσεις και από άλλους τομείς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο στον κανονισμό του EIT προβλέπεται η δημιουργία του Ιδρύματος EIT που έχει έναν μοναδικό στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο. Σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση δεν μπορώ να σας πω από τώρα το τι θα κάνουμε. Πρώτα θα πρέπει να αποφασίσουμε για το ποιους τομείς θα καλύψουμε, σε ποιους τομείς θα διευρυνθούμε και πόσα κίξ θα έχουμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ εγκαρδιότητα κύριε Επίτροπε για την επίσκεψή σα για τις πληροφορίες σα. για τις αναλυτικές σας απαντήσεις και θα ήθελα να υπενθυμίσω στην, στα μέλη της Επιτροπής στις 25 Μαΐου έχουμε το θέμα πάλι στην ημερησία διάταξη με τρεις εκπροσώπους από τα τρία ΚΙΚ θα μάθουμε δηλαδή ακόμα περισσότερα και πιο νέα γιατί είναι εν εξελίξη η διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι από τι εξελίξει. Αλλά θέλει κάτι να προσθέσει η Επίτροπο, νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι ξέχασα μια ε, ερώτηση που θα ήθελα να απαντηθεί επίσης. Όσον αφορά την ερώτηση τη κυρία Μέρκη, πώς θα συνεργαστούμε με τα EIP και με την κυρία Γιέκα Κουίν ούτως ώστε όλα αυτά να ενταχθούν σε ένα ενίο σύστημα. Είχα πάρα πολύ καλές συζητήσεις με την κυρία Κία Κουίν. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι η συνεργασία με τα ΕΕΠ που προστίθεται να εγκαθιδρύσει. Ένα υπάρχει μέχρι στιγμή όσον αφορά την ε, γύρανση, αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε συνέργειες, στο μέλλον θα το λάβουμε υπόψη μας. Έχει όμως τελείως διαφορετική μορφή <clears throat> το EIT. Η παιδεία ας πούμε είναι μια πτυχή που δεν έχει το EIP. Θα μπορούσαμε να έχουμε όμως και ένα κικ για την υγιή γύρανση Φερρυπίν. Γιατί όχι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ακόμα. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες. Αλλά όσον αφορά το EIP για την υγιή γύρανση θα μπορέσουμε να το βάλουμε στο EIT, ή στο σχετικό ΚΙΚ, για να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να εκμεταλλευόμαστε με τις εμπειρίες και τις γνώσεις των ΔΕ. Τόσο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ολοκληρώνει την εξέταση αυτού του σημείου. Τα ξαναλέμε αργότερα. Thank θα ήθελα να πάρω στο επόμενο σημείο τη ημερησίας διάταξη. Θα πρέπει να είναι το τελευταίο σημείο νομίζω. Αποζηματική στρατηγική για τι πρώτε ύλε στην Ευρώπη. Ο εισηγητή ε, συνάδελφος Κόφερ, έχει πρώτο το λόγο. Παρακαλώ. Μια εισαγωγική παρουσίαση. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ελπίζω να ανοίξουμε καλά τη συζήτηση αυτή. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Χόκμαρ και εσάς, τον ίδιο που δώσατε την εδότητα να υπάρχει αυτή η αντιστροφή των δύο σημείων στην ημερησία διάταξη για να μπορέσω να είμαι παρόν και στον τριμερή διάλογο για την διπλή χρήση, dual use. Θα ήθελα να κάνω πολύ λίγες εγωγικές παρατηρήσεις. Κατά τα άλλα, Περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τα σχόλια και επεξηγήσω των συναδέλφων. Τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να παρακαλώ το Κομισιόν να δείξει κατανόηση για κάποια διατύπωση που υπάρχει σε αυτή την πρόταση έκθεσης που δίνει την εντύπωση ότι τα υποκατάστατα δεν χρησιμοποιούνται. Ο, καθόλου δεν είναι σωστό αυτό. Μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσον λαμβάνεται αρκετά υπόψη η υποκατάσταση. Θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Δεν επιτρέπεται όμως να δίνουμε την εντύπωση του Κομισιόν ότι έχει παραβλέψει αυτό τελείως. Δεύτερον, Μία σειρά συναδέλφων υπέβαλαν κάποιε ιδέε προ. εμέ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, παραδείγματο τον Αλφα Παναγιώτοφ, ο οποίο παρουσίασε κάποιε συγκεκριμένε ιδέε που τι κατανόησα πλήρω, μου φάνηκαν πάρα πολύ σημαντικέ και ελπίζω και με άλλε παρουσιάσει συναδέλφων να έχουμε τελικά μια καλή έκθεση. Τρίτον, θα ήθελα να πω ότι έχω και εγώ κάποιε ιδέε που δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμα στο κείμενο γιατί ήταν λίγο το πρόβλημα χώρου δεν αρκούσε να αναφερθούμε σε όλα όσα θέλαμε να αναφέρουμε. η διαδικασία αυτή. Τέταρτον, η έκθεση αρχικά είχε γραφεί στα αγγλικά. Εγώ δεν έχω ελέγξει παραδείγματος χάρη το γερμανικό κείμενο τώρα. Τουλάχιστον όμως σε ένα σημείο το γερμανικό κείμενο, η γερμανική μετάφραση του αγγλικού κειμένου είναι παρεξηγήσιμη για να μην πω εσφαλμένη και θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας συγκεκριμένα. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση θα ήθελα να σας το παρουσιάσω. Στο αρχικό αγγλικό κείμενο λέει τονίζει ότι από αποτελεσματική διαχείριση της πολιτικής ε, πρώτων υλών για μία βιομηχανική ε, πολιτική, αποτελεσματική πολιτική. Ε, το γερμανικό κείμενο δεν αποδίδει ακριβώς αυτή τη σημασία και θα ήθελα παρακαλώ να κρίνετε όχι το γερμανικό αλλά το αγγλικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Θα αρχίσουμε. Καταρχήν, οι σκιώτες χιτές, ο κ. Παναγιώτοφ, πρώτος. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πατικόφερ για την τόσο καλή έκθεσή του. Η έκθεση αυτή είναι ζωτική σημασία για την Ευρώπη. Γιατί πάνω από τρία δις το χρόνο ξοδεύει η Ευρώπη για να συντηρεί τις επιχειρήσεις της, τα κομπιούτερ κτλ. κτλ με ύλες που έρχονται συνήθως από την ε, Νότια Αφρική, τον Καναδά. Αν βρείτε λοιπόν τρόπο να περικόψετε τις δαπάνες αυτές, τα χρήματα αυτά θα πηγαίνανε στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, ε, στα φάρμακα κλπ. Αν δηλαδή φροντίσουμε να ε, κάνουμε περικοπές, θα μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους ότι να έχουμε βρει τον τρόπο οποιαδήποτε κρίση στο μέλλον θα μπορέσετε να την επιλύσετε. Η έκθεση του κ. Μπατικόφερ είναι πολύ σημαντική και για έναν άλλο λόγο, γιατί αναφέρει, εντοπίζει το πρόβλημα, αλλά προτείνει και λύσεις. Για παράδειγμα, διπλωματία πρώτων υλών. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, οι υποδομές και οι πρώτες ύλε, αλλά και το know-how σε σχέση με τις πρώτες ύλε. Και γιατί. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα για νέες τεχνολογίες, έρευνα, εξοπλισμό. Ναι. Την τεχνολογία την έχει και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και σε άλλες χώρες για να λύσει και εκεί προβλήματα και να μπορέσει έτσι να προμηθεύεται πρώτες ύλες. Δύο παρατηρήσεις έχω. Πρώτον, μήπως να ξανανοίξουμε κάποια ορυχεία στην Ευρώπη. Γιατί όταν κλείνουν, όταν κλείσανε την δεκαετία του 90 τα ορυχεία, οι λόγοι ήταν διαφορετικοί οικολογική, κοινωνική, πολιτική και κυρίως οικονομική. Θυμηθείτε ότι ο χαλκός, ο τόνος τότε ήταν 1500 δολάρια αμερικανικά, ενώ τώρα είναι 10.000. Το ίδιο σχήκε για τον ψευδάργυρο, τον μόλιδο κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το ξαναδούμε αυτό και να ξανανοίξουμε κάποια ορυχεία στην Ευρώπη για να μας τροφοδετούν. Στη Βουλγαρία για παράδειγμα έχουμε για μόλιβδο, χαλκό, ε, χρυσό επίσης, υπάρχουν τέτοια ορυχεία. Θα έπρεπε να το σκεφτούμε. Και δεν ξέρω κύριε Πετικόφερ, είπατε ότι για μια περιορισμένη περίοδο κλπ. κλπ η Ευρώπη χρειάζεται μακροπρόθεσμα, όχι βραχυπρόθεσμα να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Κίνα και αλλού. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Σιμάνσκι. Ευχαριστώ για την έκθεση που μας παρουσιάσατε. Πιστεύω και εγώ ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση έχουμε πια μια καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία στην Επιτροπή μας. Ένα κείμενο το οποίο δεν είναι τόσο νομοθετικό αλλά περιγραφικό της κατάστασης έχει πολύ μεγάλη σημασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της να ισορροπεί κάπως ε, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε λίγο περισσότερο τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των τριών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με την πολιτική στον τομέα των πρώτων υλών. Το θέμα της ανακύκλωσης, την εμπορική πολιτική και την σωστή χρήση των πόρων. Δεν θα πρέπει να κάνουμε διακρίσεις εις βάρος ενός από, αυτά, από αυτούς τους τομείς, γιατί ο κάθε τομέας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε. Η χρήση των πόρων θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο υποβάλλεται θα έλεγα στους κανόνες για το σεβασμό του περιβάλλοντος και ε, φυσικά αυτό είναι το πλαίσιο, ε, το Natura 2000 είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Νομίζω ότι ότι μία άλλη προϋπόθεση ε, σημαντική είναι η ανακύκλωση και οι νέοι κανόνες αποτελεσματικότητας στον τομέα της ανακύκλωσης. θα πρέπει να υπάρξουν μελέτες ανεξάρτητες για τις επιπτώσεις αυτής της δραστηριότητας κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για το σύνολο της βιομηχανίας. Η βιομηχανία στην Ευρώπη λαμβάνει υπόψη την ανακύκλωση και κάνει πολλά στον τομέα της ανακύκλωσης και δεν νομίζω ότι το να επιβάλλει κανείς περαιτέρω προϋποθέσεις και περιορισμούς στη χρήση αυτής της μεθόδου είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Ένα άλλος ενδιαφέρον τομέας είναι η δυνατότητα ε, εκ νέου χρήσης με εναλλακτικό τρόπο των ε, των χωματερών. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, όπως ο τομέας της ε, ασφάλειας ε, της ενέργειας, θα πρέπει να μιλήσουμε και για ασφάλεια στην προμήθεια πρώτων υλών και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους στις συζητήσεις τους και στις δράσεις τους και οι υπηρεσίες της ε, νέας αυτής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είναι κάτι το οποίο είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τις διπλωματικές μας δραστηριότητες. Βέβαια υπάρχουν όρια στην ευθύνη την οποία μπορεί να αναλάβουν γιατί πάντα υπάρχουν οι εθνικές πλευρές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο πολιτικοί από τις προτάσεις που γίνονται και τότε θα καταλήξουμε στο να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Βαν Ευχαριστώ. Μαρίτος είναι σκιώδη συζητήτρια από τους σοσιαλιστές. Επειδή δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρους της και εκ μέρους της ομάδας. Και υποστηρίζω βέβαια και εγώ απόλυτα όλα αυτά που θα σας πω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ για την εξαίρετη εκθεσή σας. Υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που κάνετε. Για παράδειγμα, βελτίωση του 3% του ΕΠ. Πολύ ενδιαφέρον. Οικοδιαχείριση, οικολίζινγκ κλπ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που προτείνετε. Συμφωνούμε επίσης με τα συμπεράσματά σας για το ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το θέμα της αγοράς των πρώτων υλών χωριστά από τα λαγαθά. Δεν πρέπει μαζί να τα βλέπει όλα αυτά σε μια και την ίδια ανακοίνωση. Πρέπει να είναι χωριστό λοιπόν το θέμα των πρώτων υλών από το θέμα των αγαθών και την πρόσβασή τους στην αγορά. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες πρέπει να λάβει απόλυτα υπόψη τη συνεργασία για την ανάπτυξη και τι γίνεται στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Συμφωνούμε με τον εισηγητή για το ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πρόθεση των δικών μας πρώτων αλλά η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται όλες τις αρχές μας όσον αφορά την ε, συνοχή για την ανάπτυξη. Η εξόρυξη τώρα σαν αναπτασσόμενες χώρες πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφελούνται και οι δύο πλευρές. Η πρωτοβουλία αυτή δεν μπορεί να συνεισφέρει στην διαφθορά ή μια νέα απεικιοκρατία. Από τη δικιά μας την πλευρά και ιδιαίτερα από την πλευρά της Μαρίτας, μια που έρχεται από τη Βόρεια Σουηδία, όπου υπάρχει πολύ εξόριξη σε ορυχεία θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνατότητες εξόριξης πρώτων υλών. Μπορούμε να κάνουμε πολλά για να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Θα υποβάλουμε σχετικά τροπολογίες πάνω σε αυτό για την εκθεσή σας. Χαίρομαι πάντως που τονίζει και ο συγητής το θέμα της επάρκειας πόρων την ε, Ανακύκλωση επίσης. Είναι πράγματα που αναφέρονται στην έκθεση και συμφωνούμε απόλυτα. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα στον βορρά της Ευρώπης ώστε να υπάρξει και αηφόρος χρήση των πρώτων υλών αλλά και εξόριξη πρώτων υλών και επίσης πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο σε όλα αυτά. Θα υποβάλουμε κάποιε τροπολογίε. μη φοβόσαστε, δεν θα είναι τίποτα τρομερό. Κάποιε μικρέ αλλαγέ ζητάμε. Οι περισσότερε τροπολογίε μα είναι για να υπογραμμιστούν ακόμα περισσότερο αυτά που ήδη λέτε στην έκθεσή σα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκέρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο για την έκθεσή του. Αποτελεί η έκθεση αυτή μια πολύ καλή βάση για την τελική έκθεση. Αναφέρει πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Το τελευταίο βέβαια, εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην έκθεση αυτή γιατί το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια που η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει μέχρι στιγμής να αγνοεί τα θέματα των πρώτων υλών. Η επεξεργατική βιομηχανία δημιουργήθηκε καταρχήν με υψηλό επίπεδο πρώτων υλών και τότε υπήρχε καθυστέρηση όσον αφορά την, ε, τον κλάδο των πρώτων υλών που απαιτούν υψηλέ επενδύσεις μακροπρόθεσμες καθώς επίσης υπάρχουν και συμπληρωματικές απαιτήσει που πρέπει να πληρούνται και γι' αυτό οι κυβερνήσεις έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν. Δυστυχώς ε, δημιουργήθηκαν ε, όμιλοι ισχυροί παγκόσμια που επιβάλλουν τις δικές του απόψεις στην Κίνα παραδείγματος χάρη και έχω πάρα πολύ συγκεκριμένα σχόλια να κάνω. Καταρχήν όσον αφορά το σημείο 1 Το κεφάλαιο που αφορά την ε, στρατηγική για την ενέργεια, την πρώτη σύλληση για την ενέργεια. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε την ενέργεια, γιατί η οδήποτε πρώτη ύλη μπορεί να υπολογιστεί σαν ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε κατά νου αυτό. Και γι' αυτό θα έπρεπε ίσως να συζητήσουμε για την ενεργειακή κατανάλωση των πρώτων υλών. Και κάτι άλλο που δεν αφορά μόνο τις πρώτες ύλες, αλλά το νερό και τον αέρα επίσης. Ο αέρας. Πολύ σημαντική πρώτη ύλη. Παραδείγματος χάρη στην παραγωγή αζωτούχων ζωοτροφών και άλλων. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στην ιδέα της υποκατάστασης που είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τη στρατηγική για τις πρώτες ύλες. Και εδώ έχει κανένα κατά νου την ε, οικοδομική, ε, τον οικοδομικό κλάδο γιατί η ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία αλλάζει τώρα περνάει δηλαδή από κτίρια που κατασκευάζονται με μπετόν σε κτίρια που κατασκευάζονται με ξύλο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα για την ιδέα της υποκατάστασης. Αυτό σχετίζεται και άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και ζούμε. Βέβαια αυτό είναι κάπως πιο φιλοσοφικό το θέμα αν θέλετε. Όσον αφορά τώρα λεπτομερείς τροπολογίες, έχω αρκετές. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η έκθεση αυτή έχει, όπως σας είπα, πάρα πολύ υψηλή σημασία σε σχέση με άλλες εκθέσεις και όσον αφορά την ενέργεια, γιατί πιστεύω ότι η ενέργεια και οι προτισίες θα πρέπει να εξεταστούν από κοινού. Πρόεδρος, μία σειρά συνάδελφων έχω ζητήσει ακόμα τον λόγο. Παρακαλώ να προσπαθήσετε όλοι να έχετε κατά νου τον χρόνο. Ευχαριστώ για μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα με στρατηγικό θα έλεγα τρόπο. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια ειδικότερα για τις λεγόμενες σπάνιες γέες σε ορισμένα τέτοια υλικά η Κίνα παράγει το 97% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής και ανησυχώ για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σχετικά με τις σπάνιες γεές, βλέπουμε ότι η έκθεση αναφέρεται στον ρόλο της διπλωματίας των πρώτων υλών στις σχέσεις μας με την Λατινική Αμερική, την Ασία και ειδικά την Κίνα. Ιδιαίτερα με τις σπάνιες γεές υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στη Γρυλανδία. Έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώτες συζητήσεις. Η Γρυλανδία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι πολύ κοντά μας η κυβέρνηση έχει επιδείξει μια, ένα υψηλό πνεύμα ανεξαρτησίας τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει και μια απόφαση του Συμβουλίου για εταιρική σχέση με τη Γρυλανδία από το 2006. Η αρχική πρόταση συμπεριλάμβανε φυσικούς πόρους, εκπαίδευση κτλ. Αλλά στο τελικό προγραμματικό έγγραφο ο μόνος τομέας ήταν η εκπαίδευση. Νομίζω ότι η Γρυλανδία είναι ένας καλός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στενές σχέσεις με την Δανία. Έχουμε και αλλιευτική συμφωνία και διαπραγματευόμεθα επίσης και μια συμφωνία στον τομέα των ε, διαμαντιών. Έχει λοιπόν σημασία να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο στρατηγικός αυτός τομέας των σπάνιων γεών να ληφθεί υπόψη. Δεν θα αποφασίσω εγώ για μια κάποια συμφωνία στον τομέα αυτό. Οι Κινέζοι όμως είναι σε επαφές με τη Γρυλανδία. Η Κίνα επενδύει σοβαρότατα έχουν ε, πράγματι αγοράσει την ένταξή τους σε αγορές όπως η Αφρικανική και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει ταχύτατα. Κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε σαν συνεισηγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τις πρώτες ύλε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πέτη για μία σε βάθος έκθεση την οποία έχει προετοιμάσει και όπως είπε και η συνάδελφος Βαν Μπρέντ υπογραμμίζει ο εισηγητής αρκετά θέματα στα οποία συμφωνούμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια σωστή ανάλυση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δούμε τι συνθήκες επικρατούν και στον τομέα των λεγόμενων κρίσιμων προϊόντων Να δούμε επίσης και τι ε, παλαιά λατομεία μπορούν να γίνουν αντικείμενο επανεξέτασης έτσι ώστε να βεβαιωθούμε για τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν. Είναι ένα θέμα Ε, το οποίο πρέπει να συζητηθεί είναι το θέμα της εκ νέου χρήσης. Εδώ μιλάμε για αντικατάσταση, μιλάμε για ανακύκλωση, αλλά διαρωτώ αν η ανακύκλωση περιλαμβάνει και την επιλογή της εκ νέου χρήσης. Κάτι το οποίο εγώ βρίσκω εξίσου σημαντικό αλλά διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο θα παρατείνει την ε, διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, ενός υλικού και να συζητήσουμε επίσης εκ νέου και τη δυνατότητα ενός διαφορετικού οικονομικού προτύπου για την επιτάχυνση των ανακυκλωτικών δραστηριοτήτων. Έχει ήδη συζητηθεί αλλά θα πρέπει ο εισηγητής να επιμείνει περισσότερο στις επιλογές που υπάρχουν όχι μόνο για τα χημικά αλλά και για άλλα λεγόμενα κρίσιμα προϊόντα. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε κύριε Μπούτι Κόφερα αν είναι επιλογή στις λεγόμενες εξορίξεις επιφανείας να τεθεί ένα θέμα απαγόρευσης της χρήσης των παλαιών λατομείων γιατί εκεί βέβαια αν τεθεί αυτό το θέμα θα αυξηθεί η ανάγκη ανακύκλωσης. Κύριο Βιντάλ Κουάντρας, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μπούτικοφερ για μια εξαιρετική έκθεση και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια γύρω από τους τρεις πυλώνες της έκθεσης αυτής. Πρώτον, η διασφάλιση της δίκαιης παροχής και προμήθειας πρώτων υλών. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίσει την πολιτική της στον τομέα των προηθειών των πρώτων υλών και να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπάρχουσες δομές όπως τον ΠΟΕ ή τις διμερείς συμφωνίες αυτό θα πρέπει να γίνει εν πλήρη σεβασμό της ευθύνης που έχουμε να προωθήσουμε την αηφορία και στις χώρες εταίρους. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η, παροχή, η αηφορία στην παροχή των πρώτων υλών, στην προμήθεια συγγνώμη, των πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχουν τρία θέματα που είναι αλληλοσυνδεόμενα. Πρώτον, εδώ έχουμε να κάνουμε με την αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή ο ρόλος του ευρωπαϊκού επίπεδου θα είναι συντονιστικός και πρόταση συντονισμένων λύσεων όπως η ετήσια έκθεση για τις πρώτες ύλες που προτείνει ο εισηγητής στην παράγραφο 19. Δεύτερον, κάποιες διοικητικές διαδικασίες παραμένουν ένα σημαντικό εμπόδιο, είναι μια τροχοπέδη Μία ιδέα του λεγό, της λεγόμενης μονοαπευθυντικής θηρίδας μπορεί να λύσει το πρόβλημα και εδώ μπορώ να δεχτώ και την πρόταση του εισηγητή για την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Γεωλογικής Υπηρεσίας. Τίποτα δεν λέγεται όμως για τη μεγάλη καθυστέρηση χρονική η οποία χρειάζεται για την έκδοση ε, μιας άδειας εκμετάλλευσης. Εδώ ίσως το One Stop Shop μπορεί να αποβεί χρήσιμο υπάρχουν και άλλα θέματα περιβαλλοντικά τα οποία με οδηγούν στο τρίτο σημείο ε, που θέλω να σας θέσω προς εξέταση. Στην τελευταία συζήτηση την οποία κάναμε πολλοί συνάδελφοι υπογράμμισαν το ότι σε ορισμένες χώρες που έχουν δυνητικά ε, μεγάλη δυνατότητα παραγωγής πρώτων υλών υπάρχουν προστατευόμενες ζώνες πολύ μεγάλου εύρο. Στη δική μου χώρα την Ισπανία όπως σας έχω πει το 30% των διαθεσίμων γεών εντάσσονται στην Natura 2000. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ανοιχνεύσει την δυνατότητα να διευκολύνει κανείς κάπως τις διοικητικές διαδικασίες και να τις συνδυάσει βέβαια με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της αηφορίας στην εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων. Θα μπορούσε να συζητηθεί εδώ το θέμα μιας πιθανής ετικέτας για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται η εκμετάλλευση. Ο τρίτος πυλώνας τώρα για την ανακύκλωση λοιπά Και στη δική μου χώρα δυστυχώς στην Ισπανία η διαχείριση των αποβλήτων στην ουσία είναι οι χωματερές. Και περιβαλλοντικά και οικονομικά νομίζω ότι οι προτάσεις του εισηγητή παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ίσως αυτός ο στόχος του 3% του ΑΕΠ κατ' έτος να είναι κατά κάποιο τρόπο υπερφιλόδοξος. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η πρόταση δημιουργίας μιας κοινή μεθοδολογίας για την προσμέτρηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των πόρων. Ρούμπιχ. Δεν θα να ευχαριστήσω τον κύριο γιατί η έκθεση περιλαμβάνει κάποια κεντρικά σημεία που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καταρχήν το θέμα ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ξεχωριστά τις χρηματοπιστωτικές αγορές από τις αγορές ε, πρωτολυλών, γιατί οι αγορές πρωτολυλών έχουν δίκαιο τους εξέλιξη. Ε, πρέπει να δούμε πόσο διαφανής είναι βέβαια και πώς μπορούμε στον τομέα αυτό να εξασφαλίσουμε να μην διακυβεύεται η ε, σταθερή μακροπρόθεσμη τροφοδότηση. Η ετήσια έκθεση είναι πραγματικά σωστή προτέγγιση, νομίζω, όταν θέλουν τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν όλες τους τις γνώσεις ε, του θέματος. Και εκεί θα μπορούσε, νομίζω, η Κομισιόν να αναλάβει τον σχετικό συντονισμό. Συνέργειες φυσικά όσον αφορά τα απόβλητα ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο είναι πάρα πολύ ενέργεια, η κυρία Μέρκε θέλουμε να είμαστε πιο καινοτομικοί τη Ευρώπη, να έχουμε θέσει απασχόληση, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ευρώπη, θέλουμε η Ευρώπη να προχωρήσει λίγο. Τίθεται βέβαια και το θέμα του Natura 2000. Είναι σημαντικό το Natura 2000 και χαιρετώ, χαιρετίζω απόλυτα αυτά που τόνισε ο συνάδελφο Πουτικόφ. Δεν θα πρέπει να εργαζόμαστε ημέν αντίον των δε, αλλά μεν μαζί με του δε για να προχωρήσουμε. Μόνο εάν από κοινού προχωρήσουμε μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πρόταση των συστημάτων έγκρισης. Γιατί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κάποια πρότυπα και η Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση και ονοτομία θα πρέπει να μας βοηθήσει και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον στο 8ο πρόσχημα πλαίσιο για την έρευνα θα πρέπει να υπήρχε ένα ξεχωριστό κλάστερ πριν από τα υπόλοιπα. Είναι αλήθεια ότι στην Κίνα υπάρχουν πολλέ περισσότερε πρώτε ύλε από ό,τι σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου και θα έπρεπε να δούμε αν μπορούμε μέσω του ΠΟΕ να προχωρήσουμε, να γίνεται η κοινοποίηση μέσω της ΠΟΕ, να γίνεται ο συντονισμός μέσω της ΠΟΕ και διμερεί συμφωνίες να προωθούν τα σημεία αυτά και να τα παρουσιάσουν σε μας πιο ξεκάθαρα. Προβληματική μου φαίνεται η πρόταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση, ότι δηλαδή η έλλειψη των πρώτων υλών είναι πρόβλημα και των βιομηχανιών. Ε, βέβαια. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις θέσεις απασχόλησης, να δούμε κατά πόσον υπάρχει επαρκής τροφοδότηση, κατά πόσον διατηρείται η ενταγωστική δυνατότητα του κλάδου. Στο σημείο 7 ε, που αναφέρεται ο στόχος της αυτάρκειας ε, των πόρων, καλό είναι αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα γίνει αυτό γιατί χρειαζόμαστε καταρχήν μια βάση, μια μέθοδο καταμέτρησης αυτών των πόρων. Η μεθοδολογία υπ' αυτού θα πρέπει νομίζω να αναπτυχθεί και σίγουρα η Κομισιόν θα προσπαθήσει να δώσει τα στοιχεία το γρηγορότερα δυνατόν ούτω ώστε αυτή η αποτελεσματικότητα, η αποτελεσματική χρήση να καταμετράται. Και η συζήτηση για τους ε, Φόρος Είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε ούτως ώστε να μην διαταραχθεί η ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει, νομίζω, η δυνατότητα αφορολογικών ελαφρύνσεων και αυτά όλα αφορούν βέβαια όλο τον κόσμο, όχι μόνο την ευρωπαϊκή πλευρά. Θέλουμε δηλαδή από μια μεριά να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη, θέλουμε να αυξήσουμε την ε, δυνατότητα επενδύσεων σε κάποια επιχείρηση και αυτό σημαίνει περισσότερο κεφάλαιο και θα πρέπει στα φορολογικά θέματα να είμαστε ευέλικτοι, ώστε οι επιχειρήσει αυτές να μην βαρνηθούν, αλλά να είχαν ελαφρύσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πολύ σύντομα την Κομισιόν, ο κύριος Κουζιγκό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την Επιτροπή σας και τον κύριο Πέτη Κόφερ για τη στήριξή σας στη στρατηγική την οποία ακολουθούμε πρόσβαση στις πρώτες ύλες εκτός της Ένωσης, εντός της Ένωσης και αποτελεσματικότητα στην χρήση και η ανακύκλωση τέθηκε και το θέμα της αντικατάστασης κάποιων πρώτων υλών. Τρεις παρατηρήσεις λοιπόν. Η πρώτη αφορά την έκκληση για την εταιρική σχέση και την καινοτομία. Εμείς ε, εδώ ε, σημειώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις, δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση, αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε σύντομα για τους σπόρους τους φυσικούς που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές αρμοδιότητες ανήκουν στα κράτη-μέλη. Οπότε ε, πολλές φορές μάλιστα και σε υποεθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο δηλαδή. Οπότε εμείς δεν μπορούμε παρά να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τις πλέον χρηστές των πρακτικών. Από αυτό θα εξαρτηθεί επίσης και η επιθυμία τους ε, να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή της απλούστευσης των διαδικασιών. Ένα τελευταίο θέμα σχετικά με την Αφρική. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να προτείνουμε λύσεις win-win, δηλαδή οι πρώτες συμφωνίες τις οποίες έχουμε κάνει με την ε, Αφρικανική Ένωση ε, αφορούν και τις γεωλογικές γνώσεις και την οικονομική συνεργασία και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με νεο νεοαπικιοκρατικές τάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συγητής έχει το λόγο πάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα σύνομα να αναφερθώ σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Καταρχήν βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους θετικές ή και κριτικές. Νομίζω ότι γενικά έχουμε μια βάση ε, συνεργασίας ε, και ε, συνένεσης. Αυτό που είπε ο κ. Παναγιώτοφ όσον αφορά την μακροπρόθεσμη εξάρτηση από την Κίνα. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος γιατί τα προγνωστικά που γνωρίζω εγώ δίνουν εντύπωση ότι η Κίνα σε 10 χρόνια θα γίνει χώρα εισαγωγής λόγω της αύξησης ε, της κατανάλωσης των πρώτων υλών αυτών στην Κίνα. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην βασιστούμε πάρα πολύ ε, στην Κίνα η οποία θα μπορέσει να ικανοποιήσει μακροπρόθεσμα τις δικές μας ανάγκες. Ε, εξαρτώμεθα από την ανάπτυξη άλλων πηγών. Βέβαια, στη μαθηματική περίοδο εξαρτόμαστε από την Κίνα όσον αφορά τις παλιές χωματορές που αναφέρθηκαν. Ξέρω ότι η βιομηχανία είναι ήδη πάρα πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό. Ε, αναζητά και λέγεται παραδείγματος χάρη σε παλιές χωματερές ε, ε απορριμμάτων οικοκυριών υπάρχουν 3 με 4% μεταλλικά απορρίμματα τα οποία αξίζει πραγματικά να τύχουν εκμετάλλευση. Υπάρχουν όμως και άλλες ίσως χωματερές από βιομηχανία ή από μεταλλουργία που αξίζει ακόμα περισσότερο να χρησιμοποιηθούν. Το θέμα των πρώτων υλών όπως το έθιξε ο κύριος Σιμάσκι θα μπορούμε να έχουμε μια ασφάλεια τροφοδότησης μόνο εάν υπάρχουν ταυτόχρονα στρατηγικές ζήτησης και ε, προσφοράς. Παραδείγματος χάρη η Ιαπωνία για τις ε, σπάνιες γεές έχουν το στόχο σε 10 χρόνια να μειώσουν κατά ένα τρίτο τις ανάγκες τους στις ε, σπάνιες αυτές γεές γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν με α, συμπληρωματικές πηγές να καλύψουν τις ανάγκες τους. Λοιπόν, χρειαζόμαστε στρατηγικές ε, που θα ισορροπούν την προσφορά. Το να ληφθούν υπόψη οι πρώτε για την ενέργεια, αυτό που έθιξε ο κύριος Γκυρίκ, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάλι τίθεται το θέμα των πλεονεκτημάτων της ανακύκλωσης. Αυτό θα πρέπει πραγματικά να μην το ξεχάσουμε. Ο κύριος Μπένστεν αναφερθεί στην Γρυλανδία που σε σχέση με τον χώρο ε, της Ακτικής ε, και την ε, θάλασσα του Μπάρεντ αναφέρεται, αν δεν κλανώ στην παράγραφο 20, λέγεται ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολύ ενεργό πολιτική, ιδίω αν είναι τουλάχιστον σωστές στιγμές μου πληροφορίες, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να φροντίσουμε γιατί φαίνεται Αυστραλοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Γρυλανδία και ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Συμμερίζομαι λοιπόν την δική σας άποψη ότι δεν πρέπει να περιμένουμε στα παρασκήνια έχοντας κατ' βέβαια όλα τα σχετικά προβλήματα. Ε, ανακύκλωση, δεύτερη χρήση, όπως είπε η Σανφο Μέρκης, νομίζω ότι αν το εξτάσουμε τα πράγματα ε, συστηματικά μπορούμε η εκ νέου χρήση να θεωρηθεί σαν ένα υποκεφάλαιο της ανακύκλωσης. Για πρακτικού λόγους ήταν ίσως καλύτερο να τα αναφέρουμε και τα δύο ξεχωριστά, γιατί αλλιώ δεν θα το καταλάβουν, δεν θα το συσχετήσουν όλοι. Ναι, πραγματικά θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά. Για τι χαματορές τώρα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το προσπαθήσουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ τίνω ε, στην αρχή της επικουρικότητας την οποία ε, μας υπενθύμισε και ο κ. Βιδάλ Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν θέλω να επιβαρύνω το ευρωπαϊκό επίπεδο με έργα που μπορούν να αναλυφθούν στα πλαίσια της επικουρικότητας από τα κράτη-μέλη ή από περιφέρειες των κρατών μελών. Τι έχει το θέμα παραδείγματος χάρη κατά πόσον υπάρχουν υπερβολικά πολλές περιοχές ε, Natura 2000 στην Ισπανία. Αυτό δεν είναι θέμα που θα αποφασίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι θέμα της ισπανικής πολιτικής. Και τέλος, προς τον κύριο Ρουιμπίκ, όσον αφορά τη φορολόγηση των πρώτων υλών, ίσως εξέπληξε ορισμένους ότι εγώ δεν προτείνω γενική φορολόγηση των πρώτων Αυτό το κάνω εγνώσιμο. Υπάρχουν διάφορες ε, σκέψεις ε, στις οποίες μπορεί να βασιστεί κανένας, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι το θέμα των φόρων θα πρέπει να μελετηθεί από πλευρά στρατηγική συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι δεν πρέπει να έχουμε εδώ μια νέα συζήτηση αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων, ε, φόρων. Συγγνώμη. Α, γι' αυτό δεν θα είχε κανένα κατανόηση. Αλλά μήπως θα πρέπει εδώ πρακτικά να εξετάσουμε που θα επιβληθεί ένας φόρος, αν από την άλλη μεριά έχουμε και μία αλάφρυνση. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά σχόλια που είχα να κάνω όπου ίσως υπήρχαν ήδη κάποιες διαφορές απόψεων, από νομίζω πως θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε πάνω σε αυτές. Πρόεδρος. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτηση. Θα ήθελα να ε, σας υπενθυμίσω ότι 12 Απριλίου είναι η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. Μπορείτε να, να, να, στοιχεί, να βάλουμε στοίχημα θα είναι 500 ή 1000 τροπολογίες. Πρόεδρος. Λοιπόν, όσο το δυνατόν περισσότερες τροπολογίες να υποβάλλεται να έχει πολλή δουλειά ο κύριος Σπιτιγκόφερ Κοιτάξτε, δεν ξέρω, λόγω της ε, γερμανικής πολιτικής δεν ξέρω αν θα έχω χρόνο. Ε, αν δεν σιωπήσετε αυτή τη στιγμή θα σας γράψω εγώ πολλές τροπολογίες, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, είπαμε, το σημαντικότερο είναι η προθεσμία. 12 Απριλίου, Κατά τα άλλα θα συναντηθούμε πάλι 11 ε, ε, ε, και 13 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.